Πριν από το Συμβούλιο Μεταφορών τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο είχαμε το άτυπο Συμβούλιο της Λαροσέλου που ασχοληθήκαμε με το θέμα της ασφάλειας στη θάλασσα και μπορέσαμε να έχουμε μεγάλη πρόοδο χάρη και στη βοήθεια των κυρίων Κώστα και Σαβαρή αλλά και τη συνεισφορά του Επιτρόπου Ταγιάννη και των συνεργατών του. Έτσι μπορέσαμε όλοι να δείξουμε πόσο αποφασισμένοι είμαστε να έχουμε ευτυχή κατάληξη σε αυτό το φάκελο. Άλλοι λόγοι για τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη συνεργασία σας ήταν η συνετοχή σας σε εκδηλώσεις όπως οι μέρες ε, για τα δίκτυα τα διευρωπαϊκά μεταφορών 14 και 15 Οκτωβρίου όπου συζητήσαμε ιδιαίτερα θέματα που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή και τη χρηματοδότηση. Να πω εδώ ότι κατάλαβα πόσο αποφασισμένα είναι τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τις δεσμεύσεις τους ε, για να περάσουμε σε όλο και μεγαλύτερη διασύνδεση των δικτύων μας, ε, κάτι που αφορά και τη σύνδεσή μας με τις ε, νότιες όχθες της Μεσογείου. Σε αυτό το πλαίσιο συμμετείχαν στο άτυπο συμβούλιο και υπουργοί από τρεις χώρες του Μαγκρέμπ. Ένα άλλο σημαντικό θέμα τώρα αφορούσε τις εμπορευματικές υδροδρομικές μεταφορές και το σχετικό φόρουμ. Επίσης είχαμε την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για την Πολιτική Αεροπορία στο Μπορντό, που ασχολήθηκε με τις τεχνολογικές καινοτομίες στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος. Και εδώ είχαμε δύο σημαντικές υπογραφές. Η μία αφορούσε την πρωτοβουλία Clean Sky, καθαρός ουρανός, και η δεύτερη αφορούσε τις σχέσεις με τους παρόχους υπηρεσιών του μπλοκ της Κεντρικής Ευρώπης. Επίσης ε, είχαμε και την έναρξη του προγράμματος ΣΕΖΑΡ, κάτι πολύ σημαντικό για την επίτευξη του ενιαίου ουρανού. Είχαμε επίσης και την Ευρωπαϊκή ημέρα της οδικής ασφάλειας, όπως χαληθήκαμε και με θέματα διασυνοριακών κυρώσεων. Γενικά λοιπόν οι στόχοι μας ήταν μεταφορές ευρωπαϊκές πιο ασφαλείς, πιο καθαρές, πιο αποδοτικές και περισσότερο ολοκληρωμένες. Στα πλαίσια της ε, καταπολέμησης των κλιματικών ε, αλλαγών και μετά από το πακέτο των Υπουργών για την Ενέργεια και το Κλίμα, αλλά και σε σχέση με την οικονομική κρίση, που σημαίνει ότι μειώνονται τα περιθώρια κέρδη των επιχειρήσεων, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί πλέον υποφέρουν πολύ οι επιχειρήσεις μεταφορών. Όσον αφορά την ομοθεσία τώρα, θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα θέμα όπου είχαμε πολύ καλή συνεργασία αυτός της ασφάλειας στην θάλασσα. Κατά τη γνώμη μου ήταν ένα από τα δυνατά σημεία της Προεδρίας μας. Η πρόταση της Κομισιόν ήταν από τον Νοέμβριο του 2005 και αφορούσε δύο βασικούς άξονες, πρόληψη ατυχημάτων και μόλυνσης και συνέχεια αντιμετώπιση των ατυχημάτων. Συζητήθηκε το θέμα στο άτυπο συμβούλιο στη Λαροσέλα και παρόλο που είχε αρχικά απορριφθεί τον Απρίλιο το σχέδιο, τελικά στις 8 Δεκεμβρίου είχαμε συμφωνία στην συνδιαλλαγή και καταφέραμε τελικά να έχουμε έγκριση από το Συμβούλιο του πακέτου ΕΡΙΚΑ 3. και έτσι ολοκληρώνουμε τον κύκλο αυτό με τα δύο προηγούμενα πακέτα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για το συμβιβασμό τόσο το Κοινοβούλιο όσο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να ολοκληρώσουμε την ασφάλεια στη θάλασσα, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο κείμενα συμπληρωματικά το ψήφισμα για το κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενός συστήματος αναγνώρισης εξ αποστάσεως παρακολούθησης πλοίων του LRIT καθώς και την έγκριση της οδηγίας για την κατάρτιση των ναυτικών. Βεβαίως υπάρχει και κάτι για το οποίο λυπάμαι, θα καταλάβατε γιατί μιλάω, για το θέμα της οδικής ασφάλειας βεβαίως και για το σχέδιο οδηγίας για τις ε, διασυνοριακές οδικές κυρώσεις. Υπήρχε μεν ε, ένα κοινό πεδίο απόψεων μεταξύ Κοινοβουλίου Προεδρίας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά δεν καταφέραμε να κάνουμε αυτά που ελπίσουμε, παρόλο που εμείς θεωρούμε ότι οι κυρώσεις πρέπει να υπάρχουν, πρέπει να υπάρχει ο φόβος των κυρώσεων και αυτό πρέπει να ισχύει παντού χωρίς διακρίσεις σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Σε πολιτικό επίπεδο είχαμε συνένεση. Δεν άκουσα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας αποκλίνουσες απόψεις. Όμως, στο νομοθετικό κομμάτι δεν μπορέσαμε να έχουμε συμφωνία με τα κράτη-μέλη στα πλαίσια του πρώτου πυλώνα. Είμαστε όμοιροι, αν θέλετε, των νομοθετικών διατάξεων. Παρόλα αυτά θα ήθελα να συγχαρώ την αγαπητή κυρία Αγιάλα Σεντέρ για την πολύ ποιοτική και φιλόδοξη έκθεσή της είναι κρίμα που δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε και που σκοντάψαμε στους πυλώνες. Μία ακόμη μεγάλη πρόκληση και για εμάς αλλά και για τις επόμενες ε, προεδρίες είναι οι μεταφορές σε σχέση με την προστασία και το σεβασμό του περιβάλλοντος. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τη διάσκεψη στο Τόκιο. Ο Επίτροπος ο κύριος Σταγιάννη ήταν παρόν. Υπήρξε και η σχετική υπουργική δήλωση για την περίοδο μεταξύ Τόκιο και Κοπενχάγης. Θεωρούμε ότι στο πλαίσιο των αεροπορικών μεταφορών κάναμε ένα σημαντικό βήμα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία που εντάσσει τις αεροπορικές μεταφορές στο σύστημα ε, ανταλλαγής ε, ακπομπών αερίων. Ο στόχος είναι για εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα μειωμένες κατά 3% το 2012 και κατά 5% μέχρι το 2020 έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις διεθνείς μας υποχρεώσεις. Όσον αφορά τις οδικές μεταφορές, είχαμε το πακέτο Ταγιάννη για την μετατροπή σε οικολογικές των μεταφορών. Ασχοληθήκαμε με επίσης με το πακέτο για τις πράσινες μεταφορές. Είχαμε τις σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου. Βεβαίως όπως γνωρίζετε αυτό το θέμα χρειάζεται ομοφωνία και παρόλα αυτά, παρόλο που ήταν δύσκολο το θέμα, καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμφωνία το Δεκέμβριο στο Συμβούλιο. Είδαμε για πρώτη φορά τα κράτη-μέλη να θέλουν να αναλάβουν και το εξωτερικό κόστος ε, των μεταφορών και παράλληλα να είναι διατεθειμένα να εφαρμόσουν την αρχή όποιος μολύνει πληρώνει σε όλα τα κράτη-μέλη, λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη τις όποιες ε, γεωγραφικές και οικονομικές ε, ιδιαιτερότητες. Ασχοληθήκαμε επίσης και με την οδηγία για την Ευρωβινιέτα είχαμε το άτυπο συμβούλιο της Ρωσέλ που ασχολήθηκε με το θέμα. Επίσης 11 συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων έγιναν για το ίδιο θέμα προκειμένου να καταλήξουμε σε κάποια συνένεση για το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και για την ε, εισαγωγή ενός σχεδίου δράσης που θα έχει ως στόχο να μειώσει τα προβλήματα που προκύπτουν από το κυκλοφοριακό πρόβλημα και να δημιουργήσει μια πιο οικολογική και περιβαλλοντική ευαίσθητη κατάσταση για τις οδικές μεταφορές. Γνωρίζω πόσο σας ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Βεβαίως ε, υπήρχαν προβλήματα, είχαμε και την οικονομική κρίση, δεν μπορέσαμε να έχουμε την πρόοδο που επιθυμούσαμε, αλλά θεωρώ ότι κατά τη διάρκεια της τσεχικής προεδρίας θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα. Σας υπενθυμίζω βεβαίως ότι οι προηγούμενοι οδηγία συζητούνταν για τρία χρόνια. Σίγουρα πάντως η Γαλλία θα στηρίξει την τσεχική προεδρία. Στα πλαίσια πάντα των καθαρών μεταφορών θα ήθελα να σας μιλήσω και για την οδηγία για την προώθηση των καθαρών οχημάτων και των οχημάτων που κάνουν οικονομία ενέργειας. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους Ευρωπαίους κατασκευαστές προς αυτή την κατεύθυνση και προς την πιο γρήγορη εμπορική εκμετάλλευση των καθαρών και πιο οικονομικών αρχημάτων. Ένας ε, ακόμη πολύ σημαντικός φάκελος στα πλαίσια και της ολοκλήρωσης και της ασφάλειας και της απόδοσης και της μείωσης ε, της ε, μόλυνσης είναι ο φάκελος του ενιαίου ουρανού που απασχολεί και τον κύριο Ταγιάννη και την κυρία Μαρινέσκου. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις τεχνολογικές καινοτομίες, αλλά παράλληλα να βελτιώσουμε και την ολοκλήρωση των αεροπορικών μεταφορών, προκειμένου να μειώσουμε τις εκπομπές αεριών. Επίσης, ε, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης ε, των, ε, της αεροπορικής κίνησης, το ΣΕΖΑΡ, αποτελεί το τεχνολογικό κομμάτι του ενιαίου ουρανού. Έχουν, ξεκίνησε το πρόγραμμα αυτό και θα μπορέσουν να υπογραφούν πλέον συμφωνίες με τις υποψήφιες επιχειρήσεις. 8 Δεκεμβρίου ήταν η εγγενίαση του συστήματος ΣΕΖΑΡ. Στο νομοθετικό πλαίσιο είχαμε την τεχνική συμφωνία για την αναθεώρηση των κανονισμών που αφορούν τον ενιαίο ουρανό. Επίσης είχαμε την συζήτηση μεταξύ των φίλων από τη Βρετανία και την Ισπανία για το, αεροπόρι, για το αεροδρόμιο με του Γιβραλτάρ και θεωρούμε ότι είναι, είμαστε κοντά σε μία συμφωνία παρόλο που γνωρίζετε ότι υπάρχουν προβλήματα που έχουν να κάνουν με την κυριαρχία. Πιστεύουμε όμως ότι η Τσεχική Προεδρία θα μπορέσει να τα καταφέρει. Όσον αφορά την ε, επέκταση των αρμοδιοτήτων της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Αεροπορικής Ασφάλειας, ασχοληθήκαμε με το θέμα, αλλά δεν είχαμε αρκετό χρόνο για να μπορέσουμε να καταλήξουμε κάπου. Τέλος να πω ότι χάρη στο έργο της Σλοβανικής Προεδρίας μπορέσαμε να καταλήξουμε σε αίσιο αποτέλεσμα σε δύο θέματα που γνωρίζετε πολύ καλά. Αυτό της οδηγίας για την εναρμόνιση των φόρων αεροδρομίων καθώς ε, και τον κανονισμό για την ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης αεροπορικών εισιτηρίων. Κάτι που επιτρέπει την ε, μείωση και των φόρων των αεροδρομίων και την ε, καλύτερη κατανομή του κόστους. Και αυτό θα έχει και ιδιαίτερες συνέπειες για τις εναλλακτικές μεταφορές. Να πω επίσης ότι είχαμε διαπραγματεύσεις ε, με το Λίβανο, την Τινησία και την Αλγερία για συμφωνία για τις αεροπορικές μεταφορές, ενώ επίσης είχαμε και ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Καναδά που υπογράφηκε στις 9 Δεκεμβρίου, ενώ συνεχίζονται και διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Αυτά όσον αφορά το έργο της ε, Γαλλικής Προεδρίας στον τομέα των μεταφορών. Γενικά νομίζω ότι είχαμε πολλά καλά νέα και λιγότερες απογοητεύσεις αυτό το εξάμεινο. Και θα ήθελα να πω εδώ ότι μετά από τον κύριο Μπαρό και ο Επίτροπος Ταγιάννη ασχολήθηκε πολύ δυναμικά με τα θέματα των μεταφορών ήταν λοιπόν πραγματικά χαρά μου που μπόρεσα να συνεργαστώ με την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Κοινοβούλιο βεβαίως. Θεωρώ ότι η συνεργασία μας με το Κοινοβούλιο αλλά και το έργο του Κοινοβουλίου από μόνο του είναι πολύ ποιοτικό. Νομίζω ότι μπορέσαμε να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Εμείς από την πλευρά μας προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι ήταν δυνατό για να ανταπεξέλθουμε στις προσδοκίες σας. Θα ήθελα τώρα να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Τσεχική Προεδρία αλλά και στην επερχόμενη Σουηδική Προεδρία. Θα είμαστε βεβαίως πάντα στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Ήταν αρκετά εκτενής, αλλά αυτό συνάδει και με τα όσα καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναφέρουμε. Μία τελευταία μικρή ερώτηση ίσως να σας απευθύνω. Αναφορικά με το έργο το οποίο θα πρέπει από κοινού να πραγματοποιήσουμε μέχρι το τέλος της ε, κοινοβουλευτική θητείας. Ναι, ε, ε, τα ενία της Προεδρίας τα έχει αναλάβει η Τσεχία, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να ελπίζουμε στη συνεργασία σας και στην υποστήριξή σας για τους φακέλους και τα θέματα αυτά τα οποία έχουμε επεξεργαστεί από κοινού. Ο κ. Ζεμπόφσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητέ Ντομινίκ. Εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω εκ μέρους της ομάδας μου για την εξαιρετική σας προεδρία. Όπως είπε άλλωστε και ο πρόεδρος, ήταν μια προεδρία η οποία διακατεχόταν από το πνεύμα της ε, δικαιοσύνης και της φιλικότητας. Θα ήθελα να τονίσω δύο στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά θεωρώ, τον ναυτιλιακό πακέτο αφενός και το οποίο δεν θα είχαμε διαπραγματευτεί, δεν θα είχαμε καταφέρει να το ολοκληρώσουμε τον Μάρτιο χωρίς τη δέσμευση του Συμβουλίου. Θεωρώ ότι πραγματικά ήταν μια τεράστια επιτυχία της Γαλλικής Προεδρίας. Κατά δεύτερον, νομίζω ότι η σύνοδος αναέρειας κυκλοφορίας των Πορτό ήταν πραγματικά εξαιρετική σύνοδος. Και στην πολιτική για τις μεταφορές ε, είχε μεγάλο αντίκτυπο και ήταν καλό το γεγονός ότι μπόρεσαμε να υπογράψουμε τη σχετική συμφωνία για τον εναέριο χώρο. Θα ήθελα να αναφέρω ένα άλλο στοιχείο στο οποίο μας υποστηρίξατε. Κατά την αναθεώρηση του συστήματος ε, ETS, ε, του συστήματος εμπορίας ρήπων, δεν αλλάξαμε στοιχεία αναφορικά με τις ε, αεροπορικές μεταφορές, γιατί με, τα, με τις ρήτρες αυτές μπορούμε να επιβάλλουμε τα τέλη χωρίς να επιβαρύνουμε υπερβολικά τις ε, αεροπορικές εταιρείε, γιατί θα το δούμε αυτό το επόμενο μήνα. Θα δούμε τους επόμενους μήνες πόσο δύσκολα θα είναι η κατάσταση και θα έχουμε πλέον μια καλή βάση με την οποία θα μπορούμε, πάνω στην οποία θα μπορούμε να διαπραγματευτούμε με του Αμερικανούς ομολόγου μα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και συμφωνώ ότι είναι κρίμα που δεν καταφέραμε να σημειώσουμε επιτυχία στη διασυνοριακή δίωξη. Η κυρία Γιάλα Σέντερ και ο συνάδελφος Κορέ κατέβαλαν ε, πολύ μεγάλες προσπάθειες, αλλά τι να γίνει. Τελευταίο στοιχείο. Υπάρχουν δύο μεγάλοι φάκελοι, τους οποίους σίγουρα θα πρέπει με επιτυχία να τους κλείσουμε πριν το τέλος της θητείας. Καταρχάς το Single European Sky, ο ενιαίος ευρωπαϊκός ε, ουρανός και η οδηγία για την ΕΑΣΑ. Είναι σημαντικό να τα βλέπουμε αυτά το ένα σε εξάρτηση του άλλου. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα δύο για το περιβάλλον στον αέριο χώρο μπορούμε να εξοικονομήσουμε τριπλάσιο, τετραπλάσιο όγκο ε, ρήπων με το Single European Sky. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και για το περιβάλλον και για την οικονομία. Και το πακέτο για την μεταφορά προϊόντων. Είναι πολύ σημαντικό το πακέτο αθωτικά γκρός όπως το ονομάζουμε να μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε σε αυτή τη θητεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ασφάλεια στις οδικές μεταφορές, για την ασφάλεια και τους όρους ε, του κλάδου των μεταφορών και για την κινητικότητα στον τομέα των προϊόντων. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλούμε, όπως έχει προβλέψει άλλωστε και η Γαλλική Προεδρία, ως προηγούμενη Προεδρία να συνδράμε τη νέα Προεδρία. Νομίζω ότι Ντομινίκ, εσύ ως Υπουργός Μεταφόρων έχεις ε, μεγάλη ορμή και μπορείς να βοηθήσεις και τους τσέχους ομολόγους σου για την επιτυχία, για να κλείσουν αυτοί οι δύο φάκελοι πριν το τέλος της θητείας. Well, thank σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον ε, Προεδρεύοντα για την εργασία του επί Γαλλικής Προεδρίας και ε, για την, ε, τον απολογισμό που έκανε σήμερα προς την Επιτροπή. Νομίζω ότι υπήρξαν κάποιες επιτυχίες και αυτό σίγουρα θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε κυρίως στον, στον πακέτο, όπου πρόκειτο για μια ε, μακροχρόνια διαδικασία που στο τέλος νομίζω ότι ε, έληξε αίσια. Και νομίζω ότι η Γαλλική Προεδρία πραγματικά εργάστηκε πολύ σκληρά ε, για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω ότι θα θυμάμαι για πολύ καιρό ε, την γαλλική μόνιμη αντιπροσωπεία με την οποία συνθήκαμε πολλές φορές. Και νομίζω ότι ε, ο, ο Γάλλος μόνος αντιπρόσωπος χαμογέλασε μόνο στο τέλος. Ε, τότε κατάλαβα ότι είχαμε σημειώσει πραγματική πρόοδο. Όταν είδα έτσι να γελάει, να χαμογελάει κάπως ο, ε, ο πρέσβης, κατάλαβα ότι κάτι κάναμε. Νομίζω πάντως ότι κατέβαλαν οι σημαντικές προσπάθειες έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Ε, κάτι το οποίο το χρειαζόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερα και το χρειαζόταν και ο ναυτιλιακός τομέας και πραγματικά αξίζεται συγχαρητήρια για αυτό το θέμα. Επίσης, όπως αναφέρατε και εσείς, ε, ε, το, το ETS, το οποίο ε, το κληρονομήσατε από την ε, Σλοβενική Προεδρία. Ε, νομίζω όμως ότι στο τέλος καταλήξαμε σε μια, ισο... σε μια ισόρροπη ρύθμιση όσον αφορά το σύστημα εμπορίας ρήπων. Στην αρχή φοβόμασταν ότι δεν θα ήταν, δεν χαρακτηριζόταν από ισορροπία είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση. Αλλά χάρη στις ικανότητές σας καταλήξαμε σε ένα σύστημα εμπορίας ρήπων που να χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ισορροπία. Ε, και όσον αφορά ε, τα οχήματα, ε, δεν είναι ελκυστικό ο τομέα. Ε, ο των μικρών οχημάτων δεν πρόκειται για μεγάλα αεροσκάφη αλλά, ή για, μεγάλα πλοία, αλλά αποτελούν μέρο τη καθημερινή μα ζωή. Και αν κανεί δει το θέμα περιβάλλον και μεταφορέ, που έθεσε ως προτεραιότητα ευθύ εξ αρχή η Γαλλική Προεδρία. Νομίζω θα καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι το θέμα και σα συν, ε, ε, συγχαίρουμε και στο θέμα αυτό. Σαν αφορά τα τέλη αεροδρομίων, και εδώ ε, είχαμε μια επιτυχία. Ξεκίνησε με μια άλλη προεδρία, αλλά το προχωρήσατε και εσείς η Γαλλική Προεδρία. Αυτές όλε τι επιτυχίε πρέπει να τι τονίσουμε και να σα συγχαρούμε. Υπάρχουν όμω και ορισμένα σημεία απογοήτευση και φαντάζομαι ότι δεν σας εκπλήρει το γεγονός αυτό, το γεγονός ότι τα αναφέρω εγώ και εσείς τα κάνατε μία ανοίξη. Στις, ε, όσον αφορά τις ε, ε διασυνοριακές ε, ε, χρηματικ... ε, ποινές στις οδικές μεταφορές. Ε, κυρίως να το συνδέσουμε το θέμα με την ασφάλεια των δρόμων και με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε και τα οποία δεν αφορούν αυτές καθεαυτές τις μεταφορές, αλλά είναι νομικής φύσεως προβλήματα. Ο καλός φίλος ο κύριος ε, Γιαζερμπόφσκι είναι δικηγόρος και ε, θα καταλάβει θέλω να πω. Κοιτάξτε, ε, υπερβολικά πολλοί δικηγόροι ανακατεύονται με τα πολιτικά ζητήματα. Θα με καταλάβει ο συνάδελφος. Έχουμε και εδώ ένα κλασικό παράδειγμα. Και όχι αρκετοί δάσκαλοι και καθηγητές. Όχι, λυπάμαι. Τέλο πάντων, αυτό το σημείο μα δημιουργεί απογοήτευση και νομίζω ότι και σε εσά δημιουργεί απογοήτευση. Τώρα, τρει πολύ σύντομε παρατηρήσει. Όσον αφορά το CRS, έχετε δίκιο. Ε, ξεπερδέψαμε κάπως, αλλά περιμένουμε την Επιτροπή ε, να εκπληρώσει τις υποσχέσεις της. Είχε πει ότι θα επανέλθει ε, στο θέμα αυτό. Γιατί ορισμένοι από εμά εξακολουθούμε να έχουμε ε, ανησυχίες όσον αφορά την, όσον αφορά, την ευθύνη των μεταφορέων για το σύστημα ηλεκτρονικών κρατήσεων. Επίσης, ε, το πρόβλημα πρόσβαση στις ε, μεταφορές, στις υποδομές. Αιώνιο πρόβλημα. Και ξέρετε ότι πολλές φορές ε, επικρίνεται και η Γαλλία γιατί δεν ανοίγει το σύστημα των συνδρομικών της ε, υποδομών ε, προς τα άλλα κράτη-μέλη. Και από άποψη συνδρομών είναι κεντρικής σημασίας η θέση της Γαλλίας. Ελπίζω λοιπόν και εδώ να υπάρξει μια κάποια κίνηση και σε εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο Γαλλίας, αλλά και σε διεθνές επίπεδο για να πετύχουμε αυτή την διαλειτουργικότητα των ε, σιδηροδρόμων και να μπορέσουμε ε, να αξιοποιούμε τις ειδομικές μεταφορές ε, με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Και τέλος αφορά το ΣΕΖΑΡ. και εδώ θέλω να πω το εξή. Και αυτό δεν αφορά μόνο τη Γαλλία αλλά και τις άλλες χώρες εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή, εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Έχετε δίκιο, πρόεδρε, ε, Προεδρεύοντα, όσον αφορά το τι μπορεί να γίνει από τα ΣΕΖΑΡ και σε επίπεδο περιβάλλοντος, αλλά εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με ε, ε τον εναέριο χώρο, ε, με την, ε, με την στρατιωτική χρήση. Και εδώ πραγματικά ε, ε, σε ορισμένες ε, περιπτώσεις χρησιμοποιείται πολύ μεγάλο μέρος του χώρου αυτού από τους ερωτικούς αποκλειστικά ενώ πολλές φορές δεν το χρειάζονται και θα μπορούσαμε να τον αξιοποιήσουμε και εμείς για ταχύτερες μεταφορές και για μείωση των εκπομπών. Αναφέρομαι λοιπόν και στο σημείο αυτό και το λέω εδώ και καιρό. Μεγάλο μέρος ε, ε, ε, καλύπτουν οι στρατιωτικές μεταφορές και ο στρατιωτικός τομέας. Πάντως σας ευχαριστούμε και εσάς και τους ε, συμβούλους σας και τους υπαλλήλους της δημόσιας διοίκησης και εργαστήκατε σκληρά και πιστέψτε με, δεν το λέω αυτό σε πολλές προεδρίες. Ευχαριστώ. Κύριε Τέρξ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Τέρξ. Να σας ευχαριστήσω και εγώ, κύριε Υπουργέ το γεγονός ότι βρίσκεστε εδώ εκ των υστέρων μετά την προεδρία σας ε, με κάνει να σκεφτώ ότι κατά την προετοιμασία πραγματικά εργαστήκατε ολόκληρους μήνες πριν ξεκινήσει η προεδρία σας για να προετοιμάσετε τους φακέλους τους οποίους ξέρατε ότι θα χρειαστεί να επεξεργαστείτε. Νομίζω ότι ο τρόπος αυτός ε, συνεργασίας με το Κοινοβούλιο ήταν πραγματικά επιτυχής και θα ήθελα να σας ξαναευχαριστήσω. Ήταν πάρα πολύ καλή η Προεδρία και σε ό,τι αφορά το επίπεδο αυτό, σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μας. Δεν θέλω να πω φυσικά ότι δεν είχαμε διαφωνίες ε, για το αντικείμενο, αλλά καταφέραμε να πετύχουμε πολλά. Οι συνάδελφοι ανέφεραν ήδη πάρα πολλά θέματα, δεν πρόκειται να τα επαναλάβω, αλλά θα ήθελα να τονίσω ένα στοιχείο, την ναυτιλιακή ασφάλεια, το τρίτο πακέτο, το οποίο με πολύ κόπο αλλά και νομίζω ότι τελικά και με πολύ τεχνική ευστάθεια εδώ στις Βρυξέλλες και στο Παρίσι καταφέρουμε να το ολοκληρώσουμε. Αν κοιτάξουμε το σύνολο που ξεκίνησε το 1994 με το Έρικα, όπου ξεκίνησε η κυρία Ντεπάτσια και τα όλα τα υπόλοιπα που ακολούθησαν στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καλύψει ένα μακρύ δρόμο, λογικό, λογική συνέπεια το ένα του άλλου. Ε, το Κοινοβούλιο διατραμάτισε το ρόλο του σε συνεργασία και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Συμβούλιο προκειμένου να διατηρήσει, αν θέλετε, την ευρωπαϊκή διάσταση και νομίζω ότι τόσο το Συμβούλιο όσο και το Κοινοβούλιο μπορούν να είναι περήφανοι για το έργο τους. Κρίμα για την ε, οδική ασφάλεια, όπως είπατε. Δεν κάναμε το βήμα που θα έπρεπε να έχουμε κάνει. Τι να γίνει όμως, αναβλήθηκε, δεν ε, χάθηκε. Το θέμα θα επανέλθει στο Συμβούλιο και τουλάχιστον θα έχουμε κάνει ήδη πολλή δουλειά για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το πακέτο αυτό. Θα ήθελα να κοιτάξω και λίγο και στο μέλλον. Γιατί τόσο το πακέτο Έρικα όσο και το θέμα της κυρίας Αγέλα Σέντερα αποδεικνύει ότι στο θέμα των οδικών μεταφορών αυτό το εθνικό ένστικτο αν θέλετε εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ κρίσιμο και πολλές, σε πολλές περιπτώσεις πολλά κράτη διστάζουν να ανοίξουν τέτοια εθνικά ζητήματα για τις μεταφορές, ότι διστάζουν να μπλεχτούν σε συνεργασία με άλλες χώρες. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και πολύ φοβάμαι ότι με την οικονομική κρίση, την οποία ανέφερε χθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα είναι πιο βαθιά από ό,τι φοβόμαστε, έχω την, ε, φοβάμαι ότι θα χειροτερεύσει η κατάσταση. Το συζητήσαμε και στους συντονιστές για το θέμα των διευρωπαϊκών δικτύων. Πρέπει να το τονίσουμε και να το ξανατονίσουμε αυτό. Η σημασία της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, τη διατήρηση των επαφών, της ε, εσωτερικής αγοράς. Νομίζω ότι και στις μεταφορές θα πρέπει να τονίσουμε όλα αυτά και ξέρω ότι είμαι στην μειονότητα. Είμαι μέρος μιας μειονότητας ε, στο Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά το καμποτάζ ελπίζω στον φάκελο της ε, βιωσιμότητας, όταν θα συζητήσουμε και τις εκθέσεις του κυρίου Γιαζεμπόφης και του κυρίου Κατράου, να μην ξεχάσουμε και αυτά τα στοιχεία. Τα επόμενα χρόνια, Πρόεδρε, θεωρώ ότι θα είναι πολύ σημαντικό να τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη και θα ζητήσω από τον Υπουργό να συνεχίσει να τα συμβάλλει αυτά στο Συμβούλιο, γιατί η δική σας η χώρα έχει αυτό το ένστικτο, το εθνικό αν θέλετε, της εθνικής προστασίας λίγο πιο έντονο από ό,τι άλλο. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. go ahead. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο πρώτα στον κύριο Κράμερ. Ε, όποιος από τους δυο σας. Όχι, στο, στον κύριο Λίχτεμπεργεν. Στην κυρία Λίχτεμπεργεν. Όποιο θέλετε. Όχι, όχι, στον κύριο Κράμερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της ομάδας μου για την παρουσίασή σας αυτή που ήταν πάρα πολύ εκτενής και το ναυτιλικό πακέτο αναφέρθηκε ήδη. Ήταν πραγματικά τεράστια η προσπάθεια και εγώ να σας απευθύνω επένους. Χωρίς τη δέσμευσή σας δεν θα το είχαμε καταφέρει να περάσουν από το πακέτο του τελευταίες δύο εκθέσεις. Ήμασταν όλοι μάλλον διστακτικοί. Άρα, για εσάς λοιπόν άξιζε τον κόπο η Προεδρία σας γιατί περάσατε αυτά τα δύο θέματα, τα άλλα ζητήματα που αναφέρθηκαν. Ε, με βρίσκουν μάλλον επιφυλεκτικό για τις αδιασυνοριακές κυρώσεις, το γεγονός ότι αυτό δεν επιτεύχθηκε. Τι γίνεται. Βλέπουμε Γάλλους ε, οι πολίτες με το πεζό τους, το ρενό τους ή και με γερμανικό αυτοκίνητο να κάνουν παραβάσεις στο μέρος του, στο Βερολίνο, χωρίς ποτέ να παίρνουν κλίση. Δεν είναι δίκαιο και δεν προωθεί και την καλαγερμανική φιλία. Γιατί ο Γάλλος πολίτης ε, δεν ε, πρόκειται να διωχθεί. Ή ο Γερμανός, ο οποίος ζει στο Λονδίνο και δεν πληρώνει το τέλος συμφόρησης και μπαίνει στο κέντρο χωρίς να πληρώνει. Όλα αυτά δεν ταιριάζουν με το ευρωπαϊκό πνεύμα. Είναι πραγματικά κομμάτια που έχουν ε, εναπομείνει πλέον παροχημένα της εθνικής πολιτικής και όλα τα αναμικά προβλήματα που προκύπτουν, ούτε αυτά είναι δυνατόν να παραμείνουν γιατί βλάπτουν την νομική βεβαιότητα. Να σας παρακαλέσω λοιπόν να συνεχίσετε να παρακολουθείτε το θέμα αυτό ακόμα και αν δεν είστε πλέον στην Προεδρία για να μην υπάρχει ούτε καν ε, περιορισμός, να μην υπάρχει ανόφλη για λόγους αρχής για να είμαστε σίγουροι ότι κανείς δεν μπορεί να είναι πάνω από τους οδικούς κανόνες. Δεύτερο θέμα που ήθελα να αναφέρω η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία ήδη από τη δεκαετία του 90 ε, δεσμεύτηκε μέχρι το 2008 να μειώσει σε 140 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο τους ρήπους. Όταν διαπίστωσαν το 2006 ότι δεν πρόκειται να το διαπιστώσουν, ε, ότι δεν πρόκειται να το πετύχουν το ποσοστό αυτό, είπαν εντάξει να πούμε μέχρι το 2012 120 γραμμάρια η γερμανική αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο είπε ότι δεν είναι δυνατόν αυτό. Παρά το γεγονός ότι η κυρία Μέρκελ στην κλιματική συζήτηση είπε ότι α, δεν, είναι αυτό, δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Άρα αναβάλαμε την επιτέξη του στόχου αυτού για το 2015 και είναι κρίμα γιατί η αυτοκινητοβιομηχανία δεν χρησιμοποίησε όσα μέσα είχε και απλά χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά ως δικαιολογία για να συνεχίζει να κοιμάται. Αυτό φυσικά δεν μπορώ να το θεωρώ ως δική σας ευθύνη, αλλά πραγματικά πρόκειται για μια ήττα της Ευρώπης. Τρίτο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω, το σύστημα εμπορίας ρήπο, το κύριο του ETS και έφυγε και ο κ. Γεζεμπόφσκι δυστυχώς. Είναι πολύ σημαντικό μίλησε για την επιπρόσθετη επιβάρυνση ε, από τις αερομεταφορές. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το θέμα. Πηγαίνοντα με το τρένο από το Βερολίνο στις Βρυξέλλες, πληρώνω ΦΠΑ 19%. Όταν παίρνω το ε, αεροπλάνο, δεν το πληρώνω αυτό το ΦΠΑ. Δεν είναι δίκαιο αυτό και δεν έχει να κάνει μόνο με την ε, μόνο με την περιβαλλοντική διάσταση, γιατί ξέρουμε ότι η ρήπανση στη στρατόσφαιρα είναι πολύ πιο ε, επικίνδυνη από ότι στην ατμόσφαιρα. Γιατί να επιτραπεί αυτή η προνομική κατάσταση δεν καταλαβαίνω. Πραγματικά λοιπόν πρέπει να καταργήσουμε τα επιπλέον προνόμια γιατί ακόμα και στη Γερμανία και στη Γαλλία ακόμα και ο σιδηρόδρομος πρέπει να πληρώνουν και αναγκάζονται να πληρώνουν τέλη ηλεκτρισμού. Και κάθε χρόνο μας ε, λείπουν κονδύλια για τον εξυγχρονισμό των συστημάτων μας. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ και αυτό το θέμα, παρόλο που δεν έχετε πλέον την Προεδρία, να συνεχίζετε να τον παρακολουθείτε προκειμένου να δημιουργηθεί τουλάχιστον μια δίκαιη κατάσταση. Κατά τα άλλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προεδρία σας και εξ ονόματος της ομάδας μου. Κύριο Ζήλεχ, το λόγο. Uh, να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο για... και την Υπουργό για τις προσπάθειες που κατέβαλε για την οδική ασφάλεια, για παράδειγμα για την αέρια τώρα κυκλοφορία. Ξέρω ότι η Γαλλική πρέτρια. είχε επενδύσει πάρα πολλά στο θέμα αυτό. Βρέθηκε μια καλή λύση και οι αεροπορικές εταιρείες ε, μπόρεσαν να συνεχίσουν να αναπτύσσονται και οι σχετικές εκθέσεις ήταν πολύ επιτυχημένες. Νομίζω ότι και η Σλοβενική Προεδρία και η Γαλλική Προεδρία κατέβαλαν ε, μεγάλους, μεγάλη προσπάθεια. Νομίζω ότι το σύστημα των κυρώσεων δεν, θα, δεν λειτουργεί ουσιαστικά, αλλά δεν θα πρέπει να χάσουμε την αισιοδοξία μας. Μπορούμε και στα πλαίσια της συνθήκης Λισαβόνας να βρούμε μια καλή λύση, να το επιλύσουμε ίσως νομικά το θέμα, αν δεν καταφέρουμε να το λύσουμε αλλιώς και να ξεπεράσουν το πρόβλημα του πρώτου πυλώνου για την τσεχική τώρα προεδρία. Θα ήθελα όπως και ο κύριος Γεζεμπόσκι να τονίσω ότι η πολιτική κατάσταση και η οικονομική κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη κατά τη Γαλλική Προεδρία. Παρ' όλα αυτά όμως το θέμα των πράσινων μεταφορών είναι πάρα πολύ σημαντικό και μάλιστα έχουμε βιώσιμους ε, σκοπούς θα πρέπει μακροπρόθεσμα να δρούμε. Λοιπόν, ε, κοιτάξτε, ε, σας άφησα να πάρετε το χρόνο, ε, αλλά, ε, το, λόγο, αλλά κοιτάξτε, δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μα. Πρέπει να δώσουμε και ε, τη δυνατότητα στον Υπουργό να απαντήσει. Λοιπόν, στου επόμενου τέσσερι συναδέλφου, σα παρακαλώ κάντε πολύ συγκεκριμένε παρατηρήσει διάρκεια ενό λεπτού. Δεν θα προλάβουμε. Κύριο Κύρκο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε ε, για την νέα Προεδρία με τους εκπροσώπους ε, της ε, Τσεχικής Δημοκρατίας. Θα ήθελα να πω πολύ σύντομα ότι πιστεύω ότι η Προεδρία της Γαλλίας ήταν πολύ καλή. Βεβαίω υπάρχουν ορισμένα τελή θέματα και εγώ θα ήθελα για τα υπόλοιπα 35 δευτερόλεπτα να σταθώ σε αυτά τα ατελή ζητήματα τα οποία αφορούν τη δική μου έκθεση ε, για ε, τα CRS ε, και πρέπει για το σύστημα εμπορίας, για το σύστημα ηλεκτρονικών κρατήσεων. Και θα ήθελα να πω το εξή, ότι ναι, είχαμε καλή συνεργασία και τώρα είμαστε σε θέση ε, ε όπου ε, ε, ενέκρινε το Συμβούλιο το ζήτημα αυτό σημείο Α. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια προθυμία για ένα χρονοδιάγραμμα ε, που θα ασχοληθεί με το θέμα του μεταφορέα και με την επίσημη ανακοίνωση, κοινοποίηση. λοιπόν, με βάση τα τελεία αυτά ζητήματα, τα ζητήματα τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί, θα ήθελα να υπάρξει συγκεκριμένη προσοχή έτσι ώστε να δράσουμε απευθείας. ο επόμενος ε, ομιλητής, ο κύριος Τεσενέ. Πολύ σύντομα λοιπόν, μάλιστα, ε, συμπληρώνοντας το συνάδελφο Σίμψον, εγώ θα ήθελα μία διευκρίνηση όσον αφορά την Ευρωβινιέτα. Γιατί πράγματι στις 9 Δεκεμβρίου δεν υπήρξε συνένεση από τη συνεδρία του Συμβουλίου και εδώ νομίζω ότι υπάρχει συλλογική ευθύνη αλλά και ευθύνη της Προεδρίας ε, και λυπάμαι. Δεύτερον, όσον αφορά την εσωτερική αγορά και το πακέτο για τι οδικέ μεταφορέ, η Εθνική Ομοσπονδία Οδικών Μεταφορών στη Γαλλία ζητεί ε, να εφαρμοστεί η ρήτρα διασφάλιση. Ε, ε, ξέρετε τη του, θέση του Υπουργού. Λοιπόν, όσον αφορά την, τη διαδικασία συνδιαλλαγή και τα αναυτιδιακά, πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό και τέλο ευχαριστούμε τον Υπουργό για ε, αυτά τα οποία είπε. Τα είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ε, συ, ε, συγχαρήκατε το Κοινοβούλιο ε, για την συμβολή μας. Μα και εμείς σας ευχαριστούμε και ευχαριστούμε και τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας για την βούληση που επέδειξε. Ο επόμενος ομιλητής. Μάλιστα, πολύ σύντομα. Ε, συγχαρητήρια. Η Γαλλική Προεδρία ήταν εξαιρετική τόσο σε απογενική άποψη, ε, ε δείξατε ηγετικό πνεύμα, αλλά και όσον αφορά τι μεταφορέ συγκεκριμένα. Χωρί αμφιβολία το ναυτιλιακό πακέτο εστέφθηκε από ιδιαίτερη επιτυχία. Δείξατε ε, ηγετική, ηγετικά χαρίσματα, πολιτική βούληση, δέσμευση υπέρ τη Ευρώπη. Μια κάποια απογοήτευση ε, όσον αφορά ε, τα διασυνοριακά ζητήματα ε, και κυρίως το θέμα των πυρηναίων. Και επίση όσον αφορά τον ενιαίο, ε, του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού, μην ανησυχείτε. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισπανία 300 χρόνια συζητάνε από τη συνθήκη του τρέχτης θέματα τα οποία μας αφορούν. Αλλά ε, καταφέρνουμε να βρούμε μια λύση. Οπότε κοιτάξτε, ε, ε, δεν, είναι, δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα εμποδίσουμε να υπάρξει πρόοδο σε συγκεκριμένο ζήτημα. Ευχαριστώ. Κυρία Ντεβιράκ. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για τις επιτυχίες της Γαλλικής Προεδρίας ε, στον τομέα των μεταφορών. Δεν θα αναφέρω ξανά όλα αυτά τα θέματα, αλλά σίγουρα πριν από λίγο καιρό κανένας δεν περίμενε ότι θα καταλήγαμε σε συμφωνία στο τρίτο πακέτο για, τις, ε, για τα ναυτιλιακά. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω για το Σεζάρα και για το δεύτερο πακέτο για τον ενιαίο ουρανό. Μας είπατε ότι υπάρχει πρόβλημα με το αεροδρόμιο του Γιβραλτάρ. Πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε πρόοδο κατά τη διάρκεια της νέας προεδρίας και συμφωνία μέχρι το επόμενο Συμβούλιο Μεταφορών. Ευχαριστώ κύριος Φερνάντες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Υπουργέ, και εγώ ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Γαλλική Προεδρία για τα αποτελέσματα στα οποία ε, κατέληξε. Ε, αποτελέσματα τα οποία ωφελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα τους Ευρωπαίους πολίτες. Θα ήθελα να σας μιλήσω για το ναυτιλιακό πακέτο. Συνάδελφοι, οι συνάδελφοι προηγούμενοι από μένα αναφέρθηκαν στο ζήτημα αυτό και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τη Γαλλική Προεδρία και εσάς συγκεκριμένα κύριε Υπουργέ, γιατί πρέπει να σας πω ότι ήμουν εισηγητής ε, ε, στο θέμα ε, των υποχρεώσεων των κρατών σημαία και θα ήθελα να υποστηρίξω τα θετικά σημεία του θέματος και της έκθεσης. και θα πρέπει να υπάρξει άμεση συσχέτιση με το θέμα τη ασφάλεια θαλάσσιων μεταφορέ γενικότερα. Το ξαναλέω λοιπόν. Η Γαλλική Προεδρία ήταν εξαιρετική. Επέτρεψε την εξάλληψη συγκεκριμένων εμποδίων, έδωσε έμφαση στην ουσία και ελπίζω η έκθεση αυτή να επιτρέψει να υπάρξει συγκεκριμένη απάντηση στο πρόβλημα της ασφάλειας. Πράγμα που, κατά την άποψή μου, θα ε, επιδράσει θετικά, σε θα έχει θετικά ωφέλη σε κοινωνικό επίπεδο και υπέρ των ε, Ευρωπαίων πολιτών. και επίσης ε, και η έκθεση του Πρόεδρου της Επιτροπής μας είναι εξαιρετική, η σχετική έκθεση και ελπίζω λοιπόν και πιστεύω ότι όλα αυτά τα θέματα δεν θα είχαν ολοκληρωθεί αν δεν είχε υπάρξει αυτό το πραγματικό άνοιγμα εκ μέρου τη Γαλλική Προεδρία. Σα ευχαριστούμε και σα συγχαίρουμε για άλλη μια φορά. Uh, ένα ακόμα πράγμα, μου το επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά το σύστημα εμπορία ε, ρήπων, ε, χαίρομαι για το αποτέλεσμα το οποίο υπήρξε και για τη συνολική συμφωνία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν, ότι δεν θα αναφέρω και κάτι που έχει να κάνει με τις ε, ε, άκρως απομακρυσμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που και αυτές είναι σημαντικές και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ε, καταβάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή. Γιατί ε, Πάντω είναι σημαντικό ότι φτάσαμε στο σημείο αυτό στο οποίο φτάσαμε. Ευχαριστώ όλου του συναδέλφου που εξέφρασαν την άποψή του. Όλοι ε, ευχαριστήσαμε ε, την Γαλλική Προεδρία για την εργασία της. Και ελπίζουμε να συνεχιστούν τα καλά αποτελέσματα και στο επόμενο εξάμεινο. Σας ευχαριστούμε άλλη μια φορά και έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Merci, euh, merci, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τα πολύ φιλικά λόγια για τη χώρα μου και για την Προεδρία της Γαλλίας. Να πω καταρχάς στον αγαπητό Γκέοργ ότι σημείωσα τα όσα υπόθηκαν για τις ε, εμπορευματικές οδικές μεταφορές. Η Γαλλία συνεισέφερε στην έγκριση ορισμένων κοινών θέσεων και η Τσεχική Προεδρία νομίζω ότι μας έχει πει ότι αυτό το θέμα θα είναι στις προτεραιότητές της. Και όπως είπα και πριν, είναι κρίμα που δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε με τις διανοσυνοριακές οδικές κυρώσεις. Να ευχαριστήσω επίσης τον κύριο Σίμψον για τα λόγια του, αν και συμφωνώ με τα όσα είπατε για το Σεζάρ. Όσον αφορά για την διαλειτουργικότητα. Πολλές χώρες χρησιμοποιούν συστήματα διοδίων για τα βαρέα οχήματα. Στη Γαλλία θα ισχύσει κάτι από το 2011 πρέπει να έχουμε ενιαίο τρόπο πληρωμής, να μην κάνουμε το ίδιο λάθος που έγινε στις αρχές του 20ου αιώνα με το σιδεροδρομικό σύστημα και ο καθένας να έχει διαφορετικό σύστημα, διαφορετικές υποδομές, διαφορετικούς κανόνες ασφαλείας και διαφορετική τιμολόγηση. Όσον αφορά την απελευθέρωση των γαλλικών σιδηροδρόμων υπήρξαν ε, αρκετά ερωτήματα. Να σας πω ότι προχωρά καλά η απελευθέρωση. Στα τέλη του 2008 οι νέοι μεταφορείς, ε, κυρίως ιδιωτικοί, αντιστοιχούσαν σε περίπου 10% μερίδιο της αγοράς και θα υπάρξει και μία απολύτως ανεξάρτητη αρχή που θα διασφαλίζει την απόλυτη διαλειτουργικότητα εντός του σιδηροδρομικού δικτύου της Γαλλίας. Για τον κύριο Στέρξ, τον ευχαριστώ για τα σχόλιά του. Είναι ανοιχτή η θέση μας ε, στο θέμα των ε, οδικών μεταφορών. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο δυσχεραίνεται πολύ από την οικονομική κρίση, περισσότερο από άλλους τομείς των μεταφορών. Και λαμβάνουμε υπόψη και το σχόλιο για τη ρήτρα διασφάλισης και τη σχέση με την Γαλλία. Όντως θα συνεχίσουμε να ενδιαφερόμαστε για το θέμα των ε, διασυνοριακών οδικών κυρώσεων θα μπορούσαν να είχαν σωθεί κάποιες εκατοντάδες ζωές χάρη στην έγκριση αυτού του σχεδίου, οπότε θα συνεχίσει να μας απασχολεί. Αλλά χρειάζονται πολλές πολιτικές προσπάθειες. Ίσως όμως είναι και ένας τρόπος να αντιμετωπίσουμε και την κρίση της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Κίρσοφ, τον κύριο Τιτσένη και εσείς αναφερθήκατε στην ρήτρα διασφάλισης. Ναι, ζητήσαμε να εφαρμοστεί για τις οδικές γαλλικές μεταφορές, αλλά δεν θυμάμαι το πρώτο σας ερώτημα. Έκανα μια διαπίστωση για την Ευρωβινιέτα. Ναι, όπως είπα και πριν, θεωρώ ότι είμαστε κοντά σε μια λύση για την Ευρωβινιέτα. Υπάρχουν βεβαίως ε, κάποιες ε, πολιτικές προθεσμίες ε, στην Ευρώπη καθώς και η οικονομική κρίση που μας αναγκάζουν να πηγαίνουμε με αργό ρυθμό συνεχώς. Ελπίζω πάντως ότι θα καταλήξουμε σε λιγότερο από τρία χρόνια που είχαν χρειαστεί για την ε, πρώτη οδηγία. Για τον κύριο Πασκουάλ και τα Πυρηναία, ελπίζω ότι η υπερχόμενη Προεδρία θα διασφαλίσουν ότι θα υπάρχει και ένα τρίτο πέρασμα μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας από την Ιβυρική Χερσόνησο. Ήδη βεβαίω υπάρχει ένα μεγάλο τούνελ που ενώνει το Περπινιάν και το Μομπελιέ με την Βαρκελόνα και είναι όντως ε, μια ιστορική ευκαιρία αυτή γιατί πρέπει όλοι μαζί να συνεπάρξουμε. Τα ερωτήματα του κυρίου Ζεράκ για το Σεζάρα η Τσεχική Προεδρία θέλει να εγκριθεί το Master Plan από το Συμβούλιο Τελημαρτίου. Και ελπίζουμε ότι θα ευοδοθεί οι προσδοκίες τους. Όσον αφορά τώρα την ιστορική διαφωνία Ηνωμένου Βασιλείου και Ισπανίας για το Βιρελατάρ, ελπίζω ότι δεν θα μας εμποδίσει και ότι έστω και τελευταία στιγμή θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε λύση, κάτι που δεν καταφέραμε να κάνουμε δυστυχώς ούτε και την τελευταία στιγμή στο τελευταίο Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά, ε, Υπουργέ κύριε Μπισερό, και επειδή η ζωή συνεχίζεται, εμείς ε, Πάμε στο επόμενο θέμα της ε, ημερήσιας διάταξης, που είναι η εξέταση τροπολογιών για την οδηγία για την Ευρωβινιέτ. Ο κύριος Καντράου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πριν ξεκινήσουμε να εξετάζουμε τις τροπολογίες, θα ήθελα καταρχάς να τονίσω και να διευκρινίσω δύο ζητήματα. Καταρχάς σε ό,τι αφορά τη χρονική συγκυρία. Μαζί με τους κοιόδους συζητητές αποφασίσαμε να συνεχιστεί σήμερα η συζήτηση φυσικά, αλλά να μην ψηφίσουμε αύριο τι τροπολογίε να αναβληθεί για τι 11 ε, Φεβρουαρίου σε μία ακρόαση της ε, Επιτροπής ε, Μεταφορών. Αυτό δεν αλλάζει καθόλου την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Κάτι δεύτερο που ήθελα, κάτι άλλο που ήθελα να σας θυμίσω τη τοποθέτηση που έχουμε ή με την ε, οδηγία για το Ευρωπαϊκό Σήμα Θελών Κυκλοφορίας. Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα κράτη-μέλη, προκειμένου να αναπτύξουν στο μέλλον ένα σύστημα για την εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους μέσω ε, διοδίων. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να αποτελέσει παρά ένα βήμα. Θα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλα βήματα για να καταλήξουμε σε ένα πιο βιώσιμο σύστημα μεταφορών. Η ίδια η πρόταση προκάλεσε πολλές αντιδράσεις και από συναδέλφους στο Κοινοβούλιο και από άλλους. 530 τροπολογίες υποβλήθηκαν, εντυπωσιακό εντυπωσιακό αριθμό και καταδεικνύει ότι πρόκειται για, ένα, μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση που θα έχει σημαντικέ επιπτώσει και για τον ίδιο τον κλάδο. Θεωρώ ότι είναι καθήκον μου ως εισηγητής από όλες αυτές τις τροπολογίες να επιλέξω κάποια στοιχεία για την ε, έκθεση, κάποια στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν την ε, συνένεση του Κοινοβουλίου, την ομοφωνία του Κοινοβουλίου. Τις τελευταίες εβδομάδες νομίζω ότι έκανα με τους κοιόντες συζητητές πολλές επικοδομητικές συζητήσεις και καταλαβαίνω ότι οι θέσεις αφετηρίας φυσικά είναι πολύ διαφορετικές, αλλά πρέπει να βρούμε μια κοινή οδό τελικά για να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Και πραγματικά έχω την αίσθηση ότι κινούμαστε προς την κατεύθυνση μια συμφωνίας για κάποια σημαντικά στοιχεία της οδηγίας αυτής. Το πρώτο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω το οποίο θα πρέπει να μας βρει σύμφωνος είναι η επιλογή των εξωτερικών δαπανών που θέλουμε να εσωτερικοποιήσουμε. Η Επιτροπή πρότεινε να συμπεριλάβουμε τη συμφόρηση, τον θόρυβο και την ε, ρήπανση της ατμόσφαιρας. Πολλές τροπολογίες λάβαμε για να βγει η συμφόρηση και να περιορίσουμε το παιδί εφαρμογής αλλά και άλλοι συνάδελφοι για να διευρύνουμε το παιδί εφαρμογής, να προσθέσουμε και άλλα θέματα. Βάσει των όσων άκουσα και βάσει των ανησυχιών που άκουσα, προσπάθησα να υποβάλω μια συμβαστική πρόταση ω εξή. Διαμορφώνεται ω εξή. Καταρχά, έχω την αίσθηση ότι δεν τίθεται θέμα για τον θόρυβο και την ύπαρξη τη ατμόσφαιρα. Συζητιέται το θέμα τη συμφόρηση και υπάρχουν και σωστά επιχειρήματα, λέει ο κόσμο και δικαίω. Γιατί να υπάρχει τέλος συμφόρησης μόνο για τα φορτηγά, ενώ πολύ καλά ξέρουμε ότι τα φορτηγά μόνο εν μέρη είναι υπεύθυνα για τη συμφόρηση. Αυτό είναι πολύ δίκαιο επιχείρημα θεωρώ. Από την άλλη, αν όντω θέλουμε σε επίπεδο κράτους μέλους να αναπτυχθεί ένα σύστημα επιβολής τελών για τη συμφόρηση, ε, πρέπει να του επιτρέψουμε, να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη να ξεκινήσουν από την επιβολή τελών στα φορτηγά. Έτσι νομίζω ότι θα πρέπει να επεξεργαστούμε την, το θέμα αυτό. Είναι συζήτηση γνωστή για το αφό και την κότα. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την οδηγία ως σημείο εκκίνησης για να εντάξουμε και όλα τα υπόλοιπα οχήματα ή αντίστροφα. Νομίζω ότι από εδώ θα πρέπει να ξεκινήσουμε, αλλά να κάνουμε και τη σύνδεση με τα άλλα οχήματα οχήματα για τα οποία δεν είμαστε αρμόδιοι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ιδιωτικά οχήματα. Να διατηρήσουμε, πιστεύω, ότι πρέπει να διατηρήσουμε τον, το τέλος της συμφόρησης. Και να προβλεφθεί ενδεχομένως ένα σύστημα για άλλα οχήματα. Να γίνει ε, μια τέτοια αναφορά σε ένα σχέδιο δράσης φυσικά με σκοπό να μειώσουμε τη συμφόρηση, γιατί αυτό είναι, το, αυτός είναι ο στόχος του αλλού εγχειρήματο. Ο στόχος θα πρέπει να είναι να μειώσουμε το εξωτερικό κόστος. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο θα συμπεριλάβω στην έκθεση είναι το διοξείδιο του άνθρακα. Αλλά προτείνω να το ψηφίσουμε ξεχωριστά γιατί καταλαβαίνετε πολύ πιο δύσκολα θα πετύχουμε συμφωνία αλλά το προσθέτω ως στοιχείο πίεσης και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο για να κάνουν αυτά που έχουν ε, αναγγείλει ότι θα κάνουν σε ό,τι αφορά την ε, εναρμόνιση, σε ό,τι αφορά τους δασμούς. Όλοι συμφωνούμε ότι οι δασμοί είναι ο καλύτερος τρόπος για την εσωτερικοποίηση του διοξιδίου του άνθρακα, γιατί ξέρετε ότι υπάρχει διαφορετικό σύστημα και διαφορετικό, διαφορετική μέθοδος υπολογισμού σε κάθε κράτος μέλος για τους δασμούς. Για να αποδείξουμε επίσης πώς ε, εσωτερικοποιείται η μη το διοξίδιο του άνθρακα σε περίπτωση που επιθυμούν τα κάτι μέλη να επιβάλλουν διόδια. Αυτά λοιπόν για την ιστορικοποίηση των εξωτερικών ε, παραγόντων. Νομίζω ότι αν καταφέρουμε να συμφωνήσουμε σε αυτά θα καταπέσουν το 1 τρίτο των ε, τροπολογιών. Ένα άλλο δεύτερο σημαντικό κεφάλαιο είναι το earmarking. Όλες οι πολιτικές ομάδες εκφράζουν σαφή βούληση να συνδεθεί η εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστος με το earmarking. Να πω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα είναι πολύ σημαντικό και στις μελλοντικές συζητήσεις. Ωστόσο έχουν ε, υποβληθεί και 50 τροπολογίες περίπου για την προσαρμογή του στοιχείου αυτού. Εγώ κατέληξα σε μια πρόταση που λαμβάνει υπόψη τις απόψεις πολλών συναδέλφων και θα πρέπει να είναι σαφές ότι το earmarking για τον τομέα των μεταφορών είναι κάτι το απαραίτητο ε, σε ό,τι αφορά τη διάθεση δηλαδή την επανεπένδυση των εσόδων δεν θα πρέπει να αποτελεί αυτό σκοπό ή να είναι ένα άλλο είδος φορολογίας και για να περιοριστούν ε, οι εξωτερικοί παράγοντες του κόστου χωρίς συνέπειες. Ένα τρίτο πακέτο έχει να κάνει με τα caps, με τα πλαφόν, με τις ανώτατες τιμές. Πολλοί συνάδελφοι αναφέρουν ότι πολύ ωραία θέλουμε να συντορικοποιήσουμε το εξωτερικό κόστος, αλλά θα υπολογίσουμε με τους τύπους που προτείνονται και να υπολογίσουμε το αποτέλεσμα στην επιβάρυνση. Να το συνυπολογίσουμε. Καταλαβαίνω ότι προκειμένου να καταλήξουμε σε συμφωνία για το περίπλοκο αυτό θέμα και για λόγους διαφάνειας ότι είναι απαραίτητο να αποδεχτούμε ανώτατα όρια για λόγους σαφήνειας. Πρότεινα λοιπόν να το δούμε αυτό αποκινούμε κάποια άλλα μικρά θέματα όπως δυνατότητα σε ευαίσθητες ορεινές περιοχές να υπολογιστούν τα ειδικά κόστη, για παράδειγμα υποδομής, στο εξωτερικό κόστος, να μην χρειάζεται να επιλέξουμε το ένα από τον δύο και προτείνω και ένα πίνακα για την ατμοσφαιρική ρήπανση. Υποβλήθηκαν πολλές ε, τροπολογίες. Ο πίνακας λαμβάνει υπόψη την εισαγωγή των οχημάτων Euro 6 και των υβριδικών οχημάτων. Κάποια άλλα ίσονο σημασία σε θέματα. Πολλοί συνάδελφοι ζήτησαν να γίνει πρόταση για την διαλειτουργικότητα και για κάποια τεχνικά στοιχεία θα το υποβάλλω. Τώρα για την τομέα εφαρμογής. Θα ήθελα να πω ότι εγώ προσωπικά είμαι πολύ ευέλικτος. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Θα ήθελα να ακούσω τι έχουν να πούν οι συνάδελφοι. Δύο επιλογές έχουμε ουσιαστικά. Είτε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να επεκτείνουμε το παιδί εφαρμογή σε όλες τις διαστικές ε, μετακινήσεις, το οποίο έχει το πλεονέκτημα ότι θα έχουμε πιο πολύ εναρμόνιση, παντού θα έχουμε τους ίδιους κανόνες. Ή η δεύτερη δυνατότητα είναι να περιορίσουμε τις, ε, το πεδίο εφαρμογή στα διευρωπαϊκά δίκτυα, το οποίο θα δώσει πιο πολύ ευελιξία στα κράτη-μέλη, στη τελική ανάλυση, γιατί θα εφαρμόσουν την οδηγία αυτή στα 10, αλλά στους υπόλοιπους δρόμους μπορούν να κάνουν όλα όσα αναφέρονται εδώ ή και περισσότερα αν θέλουν. Άρα επί της αρχής εγώ θα ήμουν υπέρ της μέγιστης δυνατής εναρμόνισης, αλλά και πάλι επαναλαμβάνω ότι είμαι ανοιχτό για τις προτάσεις ε, των συναδέλφων. Τώρα, αυτό που θέλουμε να αναθέσουμε ως δουλειά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχουμε φτάσει στην τέλεια οδηγία, στο απότατο σημείο. Δεν έχουμε φτάσει στο σημείο που θα βρεθούμε ίσως σε 30 ή 40 χρόνια. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας. Ζητούμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει ποιο είναι το αποτέλεσμα του εξωτερικού κόστους και των σχετικών επιβαρύνσεων ή μήπως θα έπρεπε να περιοριστούν τα συστήματα χρονοεξαρτώμενων τελών. Θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, επίσης να διεξάγει μια καλή ανάλυση από την πρόοδο της εταιρικοποίηση των εξωτερικών του εξωτερικού κόστους για όλα τα μέσα μεταφοράς. Αυτό είναι κάτι στο οποίο επιμένουν οι συνάδελφοι και νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε καλή επισκόπηση. Και ίσως να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει σχετική νέα νομοθεσία. Να κλείσω λέγοντας ότι βάσει των συζητήσεων τους και όντες συζητητές αύριο θα υποβάλω νέο κατάλογο ψηφοφορίας που θα περιλαμβάνει και κάποιες ελαφρώς ροποιημένες συμβαστικές προτάσεις και ίσως την επόμενη εβδομάδα, την παρεπόμενη, να διοργανώσουμε νέα συνάντηση για να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία τουλάχιστον ε, πόσο είναι δυνατόν για τα μεγάλα κεφάλαια που ανέφερα. Φυσικά εξακολουθούν να υπάρχουν ε, πάρα πολλές ε, τροπολογίες τις οποίες δεν ανέφερα. Θα αναφέρω τη γνώμη μου και στον κατάλογο των ομιλιών και θα σύστηνα στους συναδέλφους να το σχολιάσουν για να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Grazie. Grazie. Εμείς ευχαριστούμε τον εισηγητή για τη δέσμευσή του ε, και να δώσουμε το λόγο στην κυρία Κόλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ως και εισηγητρίας εισηγητρία του ΕΛΚ θα ήθελα εξ ονόματος της ομάδας μου να απαντήσω σε αυτά που μας είπε ο συνάδελφος Ελ Καντράουι. Καταρχάς σας ευχαριστούμε για τις προσπάθειες σας. Έχετε δίκιο που επαναλαμβάνετε το στόχο που πρέπει να διέπει το έργο μας. Το στόχο ότι θέλουμε να συμπεριληφθεί το εξωτερικό κόστος για όλους τους τρόπους μεταφοράς. Γιατί σας ακούω να μιλάτε πολύ για τις οδικές μεταφορές. Αλλά δεν ήταν αυτός ο στόχος. Ο στόχος ήταν να εσωτερικευτεί το κόστος, το εξωτερικό κόστος για όλες τις μεταφορές. Με απότερο σκοπό να διαμορφωθεί με πιο πράσινο τρόπο η μεταφορά. Αυτό επηρεάζει και διάφορα σημεία των παρουσιάσεών σας για τις τροπολογίες. Όντως, πολλές τροπολογίες υπευλήθησαν. Αναφέρετε και λέτε ότι τόσοι πολλοί συνάδελφοι ενδιαφέρονται για τα θέματα αυτά, αλλά θα μπορούσατε να θεωρήσετε ότι Ουσιαστικά όλες αυτές οι τροπολογίες αποτελούν κριτική στην έκθεσή σας, γιατί πολλοί συνάδελφοι είχαν την αίσθηση ότι δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν την έκθεσή σας και ότι έπρεπε να αντιτυπώσουν άλλες απόψεις. Άρα θα πρέπει να ληφθεί αυτό υπόψη. Μιλάτε για προσέγγιση μεταξύ των απόψεων. Ε, βρίσκουμε ότι μπορείτε να μας προσεγγίσετε εσείς λίγο πιο πολύ γιατί ως τώρα θεωρούμε ότι σε σημαντικά σημεία είναι μάλλον απογοητευτική η εξέλιξη και ελπίζω τις επόμενες εβδομάδες να μπορέσουμε να σημειώσουμε καλύτερα αποτελέσματα, γιατί και εμείς θέλουμε να πετύχουμε ένα κοινό αποτελέσμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πιο σημαντικά τμήματα των συμβαστικών προτάσεων, τις οποίες συζητήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, δικαίως αναφέρεται ότι για το τέλος συμφόρησης μόνο για την οδική κυκλοφορία δεν υπάρχει συνένεση στο Κοινοβούλιο. Γι' αυτό και αναζητάται συμβιβασμό. Αλλά, και αυτό κινείται προς την κατεύθυνση των όσων είπε ο συνάδελφος Στέρξ, να σας προειδοποιήσω, να σας κάνω μια κριτική παρατήρηση αναφορικά με την οδό που ακολουθούμε. Γιατί στο συμβιβασμό όπως τον προτείνεται, αναφέρεται ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υποβάλουν σχέδιο δράσης. Αυτό ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Όμως, αυτό συνεπάγεται τεράστιο γραφειοκρατικό άχθος και πολλοί συνάδελφοι με έχουν πλησιάσει και μου έχουν πει ότι αυτό για τα νέα κράτη-μέλη ιδιαίτερα θα αποτελέσει τεράστιο πρόβλημα. Και συνάδελφοι οι οποίοι δυστυχώς δεν μπορούν να παραβρεθούν εδώ σήμερα, αλλά ανησυχούν ιδιαίτερα με τις προτάσεις αυτές. Και επίσης ε, προτείνεται μία εναλλακτική διατύπωση ότι μπορούν να εισηχθεί αυτό το τέλος συμφόρησης μόνο αν συμπεριληφθούν και τα ιδιωτικά οχήματα. Ξέρετε όμως πολύ καλά ότι το Συμβούλιο δεν πρόκειται ποτέ με ποτέ να συμφωνήσει με αυτό. Πότε θα το πετύχουμε λοιπόν αυτό και γι' αυτό λοιπόν ε, κρούω τον κόδωνα του κινδύνου. Προς ποια κατεύθυνση κινούμαστε. Μια τεράστια κρατία με σχέδια δράσης. Ε, πρόεδρε, δεν πρέπει να συμφωνήσει το ΕΛΚ με αυτό το στοιχείο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη του άνθρακα και σε αυτό το στοιχείο έγιναν καλές προτάσεις. σχετικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποβολή πρότασης ε, για τον ε, τέλος των καυσίμων Ας τα αφήσουμε λοιπόν τα πράγματα έτσι. Είναι σαφή έτσι ο σύνας μην τα περιπλέξουμε άλλο. Θέλουμε μια σαφή γραμμή στο σημείο αυτό. Και αυτό σημαίνει ότι ούτε αυτό το συμβιβασμό θα μπορέσουμε να τον υποστηρίξουμε. Σε ό,τι αφορά το earmarking, θα θέλαμε να ήταν λίγο πιο σαφή στην τελική διατύπωση. Σας καλούμε λοιπόν να το κάνετε λίγο πιο έντονο, γιατί μιλάμε για την πιο πράσινη διαμόρφωση του συστήματος μεταφορών. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να τονίσουμε το θέμα αυτών των επανεπενδύσεων, αλλά θα υποστηρίξουμε τη συμβαστική αυτή πρόταση, γιατί στα θέματα αυτά είναι μάλλον παραδοσιακή η διαμάχη που ακολουθεί με το Συμβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν θα σας στηρίξουμε για να είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα κάψη. Δεν κατάλαβα από την ε, παρουσίασή σας τι ακριβώς θα προτείνετε. Υποχωρείτε στο θέμα των ΚΑΠΣ να σας κάνω εγώ μια πρόταση. Ναι, όντως. Αφήστε κατά μέρο τις προτάσεις σας και αν για το τέλος συμφόρησης θα αλλάξετε το ΚΑΠ όπως ε, προτείνετε στην προηγούμενη συμβαστική, θα καταλήξουμε πραγματικά σε απαράδεκτα υψηλά, υψηλές δαπάνες χωρίς όφελος για τον κλάδο που αντιμετωπίζει πραγματικά πρόβλημα σήμερα. Ελπίζω να υποχωρήσετε στο σημείο αυτό. Και να ακολουθήσετε μια καθαρή γραμμή σε ό,τι αφορά τα κάψη. Να δούμε τι θα γίνει και στο μέλλον. Τώρα για την τιμή για την ατμοσφαιρική ρήπανση. Αυτό το υποστηρίζουμε που το τροποποιείται και για τα πιο καθαρά οχήματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα διάφορα είδη διοδίων και για τη συμφόρηση. Η συμφόρηση πραγματικά αποτελεί ένα πρόβλημα στην Ευρώπη και κάπω θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, αλλά με αποτελεσματικό τρόπο. Να δούμε λοιπόν ποιε είναι οι δυνατότητε που προτείνει και δίνει η τρέχουσα οδηγία. Αυτό να το βλέπω στη συνόλη συζήτηση αυτή που γίνεται. Πάρα πολλέ ε, δυνατότητε που προσφέρει η τρέχουσα οδηγία δεν αξιοποιούνται από τα κράτη-μέλη. Για να δούμε λοιπόν τι έχει γίνει. δυνατότητες για την αύξηση των διοδίων, προτάσεις ε, του κυρίου, της κυρίας Πατάκη, του κυρίου Μπλόκλαντ. Προς αυτήν την κατεύθυνση θέλουμε να, κοιτα... να κινηθούμε και για τα regulatory charges, για τα ρυθμιστικά τέλη. Δεν ε, συμφωνούν όλοι για το θέμα αυτό. Να δώσουμε λοιπόν απόλυτο περιθώριο δράση στα κράτη-μέλη γιατί τελικά στις αστικές περιοχές είναι που υπάρχουν πιο έντονα προβλήματα. Ας δώσουμε λοιπόν ελευθερία δράση στα κράτη-μέλη. Αν λοιπόν το κάνουμε αυτό, νομίζω ότι αυτό θα αρκεί για μας. Δεν χρειάζεται καν το τέλος ε, συμφόρησης για το πεδίο εφαρμογή. Έγιναν πολλές ε, προτάσεις που υπερβαίνουν ουσιαστικά τα αντιευρωπαϊκά δίκτυα. Πάρα πολλές και διαφορετικές διατυπώσεις ε, για τα φορτηγά, για τις σημαντικές περιοχές και περιφέρειες, πολλές προτάσεις, αλλά καμία από τις διατυπώσεις αυτής, αυτές δεν έχει σαφή ορισμό. Λοιπόν, πού θα μπλέξουμε, σε τι συζήτηση θα μπλέξουμε. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια ξεκάθαρη γραμμή, πρόκειται για μια ευρωπαϊκή γραμμή και θα πρέπει να εστιαστούμε κυρίως στις διευρωπαϊκές μεταφορές, μετακινήσεις. Ξέρουμε τι είναι τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Έχουν ένα σαφή ορισμό. Ας μην μπλέξουμε σε τελεία συζητήσεις λοιπόν. Ας περιοριστούμε σε αυτά. Τώρα, για το μέλλον. Μία γενική παρατηρήση. Πρόεδρε, συζητάμε την προσαρμογή μιας οδηγίας η οποία δεν έχει κλείσει ούτε κανένα χρόνο ύπαρξή, Διαβάζοντας σας την πρότασή σας για τα μελλοντικά βήματα, τη συμβαστική σας πρόταση για τα μελλοντικά βήματα. Τι θα γίνει, θα ξαναρχίσουμε την προσαρμογή, θα ξαναρχίσουμε την επανεξέταση. Νομίζω ότι μπλέκουμε σε μια διαδικασία η οποία δεν είναι υπεύθυνη έναντι των κρατών μελών που θα κληθούν να τα μεταφέρουν. Μου φαίνεται ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να επιμείνουμε στην εφαρμογή των όσων ήδη έχουμε, παρά να κυνηγάμε νέους στόχους. Γιατί στην περίπτωση αυτή όλα θα παραμείνουν στο χαρτί, δεν θα γίνει τίποτα πράξη. Ξέρω ότι στην προηγούμενη οδηγία κοιτάξαμε τις μελλοντικές προοπτικές σε τρεις προτάσεις. Τώρα το κάνουμε σε 25 προτάσεις. Το διευρύνουμε. Θα ήθελα να είμαστε λίγο πιο ξεκάθαροι και να επικεντρωθούμε στα πιο σημαντικά στοιχεία. Όχι να αρχίσουμε και να προγραμματίζουμε υπερβολικά πολλά πράγματα. Ας δώσουμε λίγη ασφάλεια και στα κράτη-μέλη. Τέλος, συμφωνώ σε ό,τι αφορά τη διαδικασία ε, κυρώσεων. Είχατε προτείνει να γίνει ψηφοφορία κατά τμήματα, αλλά δεν έχουμε ακόμα την τελική μορφή των συμβιβασμών και του καταλόγου ψηφοφορίας. Θα χρειαστούμε πιο πολύ χρόνο, γιατί σίγουρα θα έχουμε τροπολογίες και θα πρέπει να δούμε και τις συμβιβαστικέ ε, τροπολογίες και αυτό με, τα, με τις ε, προοπτικές, αν δεν προσαρμόσετε την ε, συμβιβαστική τροπολογία. Θα συζητήσουμε ψηφοφορία κατά τμήματα. certamente non è mio. Κοιτάξτε, ε, δεν θέλω προς Θεού να τα παρακολύσω όλα αυτά. Ε, θα αφήσουμε ε, λίγο χρόνο ε, και σας και οδησικητή να τοποθετήσω όλα αυτά. Ο κύριος Τάρξ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ για το έργο που κάνατε κύριε Σιγητή. Το έργο σας ήταν εξαιρετικό. Είναι πιο σημαντικό να έχουμε υπόψη ότι πρόκειται για ένα πρώτο βήμα σε μια συζήτηση η οποία θα πάρει χρόνο. Και νομίζω ότι θα πρέπει να θεωρήσουμε υπό το φως αυτό ε, κάποια στοιχεία, ότι δεν ε, καθορίζουμε δηλαδή λεπτομέρειες, αλλά κάνουμε ένα πρώτο βήμα. Θα ήθελα να πω καταρχάς σε δύο λόγια για την επανεπένδυση των εσόδων το τα οποία προκύπτουν από, τις, ε, από τα τέλη αυτά. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο για μένα. Γιατί αν αυτό το ρυθμίσουμε σωστά, πολλά μπορούν να γίνουν. Αν αυτό δεν ρυθμιστεί σωστά, ό,τι και να κάνουμε θα πάει χαμένο, θα πάει στράφη. Και νομίζω ότι αυτό είναι κρίσιμο και για τις συζητήσεις μας με το Συμβούλιο. Αν επιβάλλουμε δηλαδή μόνο τέλη και δεν χρησιμοποιούμε τα έσοδα για να μειώσουμε το εξωτερικό κόστος, δεν κάνουμε τίποτα. Και θεωρώ ότι ως κοινοβούλιο συμφωνώ απόλυτα και με τον εισηγητή αλλά και με την Κορίν. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο στο οποίο θα πρέπει να επιμείνουμε ως κοινοβούλιο γιατί πολύ φοβάμαι ότι εκεί θα εστιαστεί η συζήτηση με το Συμβούλιο. Είμαι πεπισμένος ότι αν κάνουμε το πρώτο βήμα σε ένα τέτοιο σύστημα χωρίς να έχουμε ρυθμίσει το ζήτημα της επανεπένδυσης όλα τα υπόλοιπα βήματα θα πάνε χαμένα. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο θα πρέπει να υποστηρίξουμε πάρα πολύ τον εισηγητή, να μειώσουμε το εξωτερικό κόστος. Αυτό θα πρέπει να αποτελεί τον απότερο στόχο. Αυτό θα πρέπει να κάνει κάθε κράτος μέλος που επιβάλλει τέλος. Να επενδύει για τη μείωση του εξωτερικού κόστους. Μόνο για τα φορτηγά, όχι απαραίτητα. Αν ε, μπορώ να περιορίσω, για παράδειγμα, σε τομέα που πλήρεται από συμφόρηση και τα ιδιωτικά οχήματα. Ε, έτσι μειώνουμε το εξωτερικό κόστος, βοηθάμε και τα φορτηγά και τα ιδιωτικά οχήματα. Δεν θα πρέπει να περιορίσουμε το πεδίο εφαρμογή, αλλά θα πρέπει και το αποτέλεσμα να συμπεριληφθεί στο κείμενο και το κάτω μέλο θα πρέπει να υποχρεούται να αποδείξει αυτή την επίδραση, αυτή την ε, απόρρια της επιβολή του κόστου πριν ακολουθήσει τα υπόλοιπα βήματα. Τώρα, η επιλογή των εξωτερικών στοιχείων. Και στην ομάδα μου διαμορφώθηκαν διαφορετικές απόψεις. Ε, το συζητήσαμε επί μακρόν και συμφωνήσαμε στη συμφόρηση με την προϋπόθεση της επανεπένδυσης, το οποίο μας φαίνεται λογικό, αλλά όχι με το διοξίδιο του άνθρακα. Για τα ΚΑΠΣ. εκτός και αν πρόκειται, επειδή πρόκειται για το πρώτο βήμα της διαδικασίας, νομίζω ότι καλύτερα να τα αφήσουμε τα πράγματα όπως τα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και συμφωνώ με την προσαρμογή του πίνακα. Η διαλειτουργικότητα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Να μην προκύψουν 100 διαφορετικά συστήματα, ένα συμβατό πρόγραμμα σε όλα τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να το απαιτήσουμε αυτό κατευθείαν τώρα, κατά την εισαγωγή του συστήματος, να είναι διαλειτουργικό. Αυτό είναι σημαντικό για την ιστορική αγορά, γιατί αλλιώς μπορεί να περιορίσει αυτό την ε, αποδοτικότητα του συστήματος για το πεδίο εφαρμογής. Επειδή ακριβώς πρόκειται για ένα πρώτο βήμα, ας ξεκινήσουμε με τα ευρωπαϊκά δίκτυα να δούμε λειτουργεί ή δεν λειτουργεί το σύστημα αναφέροντας και τις αστικές ε, περιοχές με κάποιο τρόπο. Τα υπόλοιπα θα αφήσουμε στην επικουρικότητα. Υπάρχουν πάρα πολλέ διαφορέ μεταξύ των κρατών μελών και σε ό,τι αφορά τι γεωγραφικέ καταστάσει και το καθεξή. Α κάνουμε ένα πρώτο βήμα με τα τεν και βλέπουμε. Και άμα τα πάνε καλά, αν προχωρήσει το σύστημα στα διευρωπαϊκά δίκτυα και πάλι χαρούμενοι να είμαστε για το μέλλον, για την αξιολόγηση. Και εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που λέει η Κόριν είναι σωστό. Δεν μπορούμε να κοιτάμε το επόμενο βήμα πρωτού ολοκληρώσουμε το προηγούμενο. Θα πρέπει η αξιολόγηση να είναι λίγο πιο ευρεία και θα ήθελα να κοιτάξουμε και δύο θέματα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα στο model shift για την αλλαγή δηλαδή των τρόπων μεταφοράς και κατά δεύτερον τι συνέβη και με το εξωτερικό κόστος το ίδιο. Γιατί αυτό που κάνουμε σκοπό έχει να μειώσει το εξωτερικό κόστος. Τι συνέβη λοιπόν με το εξωτερικό κόστος μετά την εφαρμογή των μέτρων που αποφασίσαμε. Γιατί αν εφαρμόσουμε ένα μέτρο, για παράδειγμα για το θόρυβο, για τη μείωση του θορύβου, αν τελικά αυξηθεί ο θόρυβος, ε, δεν καταφέραμε τίποτα επιβάλαμε ένα τέλος στο μεταφορικό κλάδο χωρίς αποτέλεσμα. Νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία λοιπόν είναι σημαντικά και νομίζω κύριε Σεγητά ότι με τις συμβαστικές που προτείνεται καλύπτουμε μεγάλο δρόμο, αλλά κάποια στοιχεία θα πρέπει να τα εξετάσουμε εκ νέου. Ο κατάλογος ψηφοφορίας θα είναι πολύ περίπλοκος θα πρέπει να λάβουμε ένα πλαίσιο από εσά στο οποίο θα εργαστούμε, γιατί θα πρέπει να δούμε αν αποδεχτούμε τις συμβαστικές προτάσεις, ποιες τροπολογίες θα χρειαστεί να ψηφίσουμε μετά. Θα είναι πάρα πολύ περίπλοκο και θα χρειαστούμε και τη συνδρομή της γραμματείας. Θα χρειαστούμε και χρόνο στις ομάδες μας για να τα κοιτάξουμε τα πράγματα αυτά. Σας ευχαριστώ όμως για όλη την προσπάθεια που έχετε καταβάλει και ελπίζω το Συμβούλιο να παραμείνει αμετακίνητο έναντι του Συμβουλίου, δεν ξέρω και πού είναι το Συμβούλιο που κάθεται, αλλά αυτό είναι το σημείο πραγματικά στο οποίο είμαστε μετακίνητοι. Αν ο σκοπός μας δεν είναι να περιορίσουμε το εξωτερικό κόστος, ε, δεν έχει νόημα να προχωρήσουμε το σύστημα αυτό. Τελεία και Παύλα. Σας ευχαριστώ. Ähm, Äh, σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Και έχει δίκιο νομίζω ότι πρόκειται για ένα θέμα του μέλλοντος. Θα πρέπει να το εξετάσουμε σε βάθος. Για όλα όσα ακούσαμε ως τώρα, να σας παρουσιάσω και τη δική μου θέση για τα μεμονωμένα θέματα, για τη διοξίδα του άνθρακα. αν θέλει να υποβάλει η Κομισιόν πρόταση εναρμόνισης, ε, ξέρω ποια, ποιοι θα είναι οι συνήθεις ύποπτοι που θα βγουν και θα πούνε ότι α, δεν μπορούμε να το συνεχίσουμε αυτό το θέμα. Γνωρίζετε άλλωστε και τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν. Και φοβάμαι κάπως ότι το όλο θέμα θα αναβληθεί πολύ απλά και δεν θα συμβεί απολύτως τίποτα. Θα ήταν πάρα πολύ κρίμα, θεωρώ. Δεύτερο σημείο η επανεπένδυση, το earmarking. Νομίζω ότι οι εμπειρίες ως τώρα με το earmarking, όπως διατυπώνεται ως τώρα, δεν είναι καθόλου κακές. Προέκυψε μια διατύπωση αρκετά σαφής και φυσικά συμφωνώ ότι αυτός θα πρέπει να είναι ο απότερος στόχος, να περιορίσουμε το εξωτερικό κόστος ασφαλώς. η εξωτερική επιβάρυνση και το εξωτερικό κόστος. Γιατί αν δεν έχουμε πετύχει το στόχο μας αυτό δεν θα έχουμε και κόστος τελικά. Πρόκειται για κάτι που καθιερώνει τις διοικητικές δομές, όπως διαπιστώσαμε στην Αυστρία τη δεκαετία του 20 και του 30. Α, τέλος πάντων, σε ένα άλλο θέμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επιβάρυνση με διοξίδιο του άνθρακα, θα έπρεπε να συμπεριληφθεί ως δυνατότητα για τα κράτη-μέλη. Υπάρχει κάτι που να μας ε, κάνει να είμαστε αντίθετοι, δεν νομίζω. Όπως ξέρετε, αυτή η ικανότητα, αυτή η δυνατότητα, συγγνώμη, χρησιμοποιείται από πάρα πολύ λίγα κράτη-μέλη. Μιλάμε για μια δυνατότητα, όχι για εισαγωγή υποχρέωση για το θέμα αυτό και για τα θέματα φυσικά είναι απαραίτητο να έχουμε ένα διαλειτουργικό σύστημα. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι δεν βλέπω να υπάρχει κάτι τέτοιο επί του παρόντος στην Ευρώπη. Δυστυχώς το διαπιστώνουμε αυτό. Θα πάρει λίγο χρόνο ακόμα, αυτό όμως αποτελεί τον απότερο στόχο. σκοπός μας δεν είναι να δημιουργήσουμε εμπόδια μέσω διαφορετικών τεχνολογικών συστημάτων, αλλά να επιλέξουμε το καλύτερο σύστημα. Και αυτό να προωθήσουμε. Να περάσουμε στα θέματα συμφόρησης. Έχουμε ένα ζήτημα αρμοδιοτήτων, γιατί πολύ απλά μπορούμε να λάβουμε ε, να προβλέψουμε διατάξεις που να μην αφορούν τα ιδιωτικά οχήματα. Το θέμα είναι πόσο θα μας βοηθήσει αυτό το να δημιουργούμε δηλαδή συστήματα τα οποία ασκούν πίεση στα κράτη-μέλη να δραστηριοποιηθούν και για τα ιδιωτικά οχήματα. Μιλάμε για τα φορτηγά, Μιλάμε για την επιβολή διοδίων για τη μείωση της συμφόρησης σε σημεία όπου όντως αποτελούν μεγάλη επιβάρυνση τα φορτηγά. Δεν είναι τόσο πολλά, είναι κάποια σημεία κλειδιά όπου τα φορτηγά παίζουν σημαντικό ρόλο. Και φυσικά υπάρχουν διαφορετικές τιμές σε διάφορους, διάφορους οδούς της Ευρώπης. Θεωρώ ότι πρόκειται για ένα θέμα Λέμε δηλαδή ότι αν υπάρχουν αυτοί οι άξονες όπου τα φορτηγά αποτελούν μεγάλη επιβάρυνση, θα σας θυμίσω κάποιους άξονες, για παράδειγμα έξω από το Μόναχο, όπου ουσιαστικά ένας δρόμος ε, είναι μονίμως γεμάτος από φορτηγά και στις Άλπεις έχουμε τέτοια προβλήματα. και δεν μπορούν καν να βγουν από τις εξόδους τα ιδιωτικά οχήματα. Αυτά θα πρέπει να τα παίρνουμε, να λάβουμε υπόψη. Υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις, δεν τις βγάζουμε από το μυαλό μας. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα της υπερβολικής συμφόρησης τώρα για τα κάψα. αν υπάρχει ένας τύπος ε, εκτίμησης και παράλληλα και ένα ανώτατο όριο και πίνακες ε, υπολογισμού, υπάρχει μία απλή λογική θεωρώ πίνακες όπου δεν υπάρχουν στοιχεία υπολογισμού και όπου ε, χρειάζεται υπολογισμός να γίνει υπολογισμός με τις, ε, τους τύπους αυτούς. Αλλιώς θα είχαμε μία τη τιμή για όλους. Δεν είναι λογικό για μένα αυτό. Γι' αυτό δεν θα ήμουν υπέρ της υποχρεωτικής διαμόρφωσης των ΚΑΠΣ. Θα το πρότεινα για τα σημεία εκείνα του πίνακα όπου δεν υπάρχουν δεδομένα. Γιατί άλλωστε είναι πάρα πολύ διαφορετικά τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη και η αντιμετώπιση τους για το θέμα αυτό σε ό,τι αφορά το σημείο εφαρμογή. Βρισκόμαστε σε μία βαθιά αντίθεση μεταξύ λογικής και ε, ρεαλισμού. Λογικό θα ήταν να συμπεριλάβουμε όσο δυνατόν πιο πολλούς τομείς, αλλά από ρεαλιστικής άποψης είναι θέμα διοδίων και θα πρέπει να πούμε ότι πολύ απλά δεν έχουμε ακόμα αυτή τη δυνατότητα. Δεν θα μπορούσαμε δηλαδή να το εφαρμόσουμε το σύστημα, ακόμη και αν συμφωνούσαμε όλοι ότι είναι η καλύτερη ιδέα θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια βαθμία προσέγγιση, αλλά ο σκοπός αυτός είναι κάτι το οποίο θα πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας. Δεν μπορούμε να παριστάνουμε ότι, ε, τι να γίνει, ο τομέας εφαρμογής ε, είναι περιορισμένο και να ξέρουμε ότι δεν πρόκειται για την ιδανική λύση. Αλλά μπορώ να φανταστώ ότι θα ξεκινήσουμε με το ΤΕΝ και μετά θα δούμε και θα αφήσουμε και περιθώριο ελεύθερε δράσεις στα κράτη-μέλη και όσο χρόνο χρειάζονται. Περιθώριο το οποίο δυστυχώς δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε. Πολλά θα είχα να αναφέρω ακόμα. Αλλά να επικεντρωθώ στα πιο σημαντικά. Ελπίζω να καταφέρουμε να διευκρινίσουμε σε κάποιες συμβιβαστικές προτάσεις ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τηρεί το λόγο του να πούμε ότι θα πρέπει να συνυπολογιστεί το εξωτερικό κόστος βαθμιαία, βαθμία, όπου δεν είναι αυτό ακόμη δυνατόν εντάξει, να προχωρήσουμε σταδιακά και κλείνοντας να πω ότι η επιβάρυνση σε κάποιους τομείς από την κυκλοφορία των φορτηγών που δεν ε, μετακινούν, δεν μεταφέρουν μόνο απαραίτητα προϊόντα από το ένα σημείο στο άλλο, είναι τεράστια η επιβάρυνση αυτή και προκύπτουν ζημιές. Προκύπτουν ζημιές, αυτό μην το ξεχνάμε. Δεν μιλάμε για παιχνίδια. Μιλάμε για περιβαλλοντικές ζημιές, για βλάβες στην υγεία, για παράγοντες ενόχλησης, για ζώνες όπου εστιάζονται όλα τα προβλήματα και για ζώνες ε, όπου δεν είναι ακόμα τόσο έντονο το πρόβλημα, αλλά θα γίνει έντονο, θα πρέπει να αντιδράσουμε. Ας ε, προβλέψουμε λοιπόν και για το μέλλον, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός. Σας απευθύνω λοιπόν έκκληση να σκεφτείτε ότι υπάρχουν και περιοχές που έχουν πολύ μεγάλη επιβάρυνση. Κοιλάδες για παράδειγμα ή ορεινές περιοχές, κάποιες ευαίσθητες περιοχές στην Ευρώπη. Το μέτρο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για τις περιοχές αυτές και όποιος θεωρεί ότι αυτό βλάπτει την οικονομία στην Ευρώπη να έχει υπόψη του ότι την προστατεύουμε την οικονομία μάλλον, την προετοιμάζουμε για το μέλλον και αυτό είναι το σημαντικό. Χρειαζόμαστε ένα έξυπνο model shift. Αυτό θα το καταφέρουμε εάν αφήσουμε κατά μέρο τους δισταγμούς, αλλά αν καταστρώνοντας σχέδια δράσης και για το μέλλον. προκειμένου να ξέρει και η οικονομία και να μπορεί να υπολογίζει πώς θα αντιμετωπίζει τα θέματα των μεταφορών. Αυτός είναι ο σκοπός μου και ελπίζω να καταφέρουμε να κάνουμε ένα πραγματικό βήμα προς τα εμπρός. Και να μην ε, επηρεαστούμε από τους λομπίστες που μας χτυπούν την πόρτα και μας ε, λένε διάφορες απίθανες ιστορίες για το ποιες θα είναι οι αρνητικές συνέπειες του μέτρου αυτού. Γιατί η εξαγωγή των προϊόντων δεν θα περιοριστεί έτσι. Αυτό το έχουμε δει άλλωστε και στο παρελθόν. Νομίζω ότι στο σημείο αυτό θα καθησυχάσουμε αρκετές από τις ανησυχίες. Ευχαριστούμε. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Τζίλε. Ναι, εκπρόσωπη των ομάδων πρώτα και μετά ε, θα δώσουμε πολύ λίγο χρόνο στους υπόλοιπους. Ε, ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κατράου για το έργο του. Γνωρίζουμε όλοι ότι βρισκόμαστε στα πρώτα βήματα και πρέπει να επιμείνουμε προκειμένου να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Όσον αφορά τον earmarking, είναι πολύ σημαντικό. Και είναι σημαντικό να καταλήξουμε σε κάποιο συμβιβασμό για το θέμα αυτό. Εμείς θα στηρίξουμε ένα συμβιβασμό. Δεν είναι πάντως εύκολο να αλλάξουμε εύκολα την ε, πρόταση της Επιτροπής ε, για τεν και για άλλες οδούς. Γιατί έχουν ε, υλοποιηθεί διαφορετικά τα τένα σε κάθε κράτος μέλος. Ακούω βεβαίω και κάποιες ε, φήμες ότι μπορεί να αλλάξει η επικρατούσα άποψη. Όσον αφορά τώρα τα ανώτερα τα όρια, δεν θεωρώ ότι είναι καλό μέτρο η άρση τους. Υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι θα ήταν ε, βλαβερές οι συνέπειες μιας άρσης ε, των ανώτατων ορίων. Πρέπει να τα κρατήσουμε λοιπόν, παρόλο που θα μπορούσαμε να έχουμε διαφορετικές ε, διατάξεις ε, για τις ορεινές περιοχές κτλ. Όσον αφορά την κυκλοφοριακή συμφόρηση, θα μπορούσαμε να έχουμε ειδικά μέτρα για τα βαρέα οχήματα κτλ. Όμως, με ανησυχούν κάποιες απόψεις και πρέπει να το δούμε τακτικά το θέμα, να δούμε πώς θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε έναν συμβιβασμό με το Συμβούλιο. Και αν καταλήξουμε σε συμβιβασμό θα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό. Σίγουρα πάντως η κυκλοφοριακή συμφόρηση είναι το πιο ακριβό κομμάτι των εξωτερικών εξόδων. Όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα τώρα. Ζητάει η Κομισιόν να συμπεριληφθεί το κόστος τους. Είναι ένα δύσκολο το θέμα αυτό αλλά και εδώ νομίζω ότι θα μπορούσαμε να βρούμε έναν συμβιβασμό. Τέλος, κάτι άλλο που αναφέρεται στη συμβιβαστική τροπολογία F αφορά ένα σύστημα με χρονικές περιόδους δεν είναι κακή ιδέα, όμως χώρες όπως η Φιλανδία, η Εστονία, η Λετωνία αν το χρησιμοποιήσουν αυτό, τότε θα αυξηθούν οι ουρές στα σύνορα των χωρών, στα σύνορα με τη Ρωσία, με την Πολωνία, για παράδειγμα. και θα υπάρχει μόλυνση σε αυτά τα σημεία τότε. Θα στηρίξω πάντως ε, εδώ την ε, πρόταση του κυρίου Κατράουη. Θεωρώ ότι αυτό αυτή η λύση με τους χρονικούς περιορισμούς δεν είναι ότι καλύτερο, αλλά σίγουρα πρόκειται για μια πολύ δύσκολη κατάσταση εδώ και εξαιρετική αν θέλετε. Ε, ε, Στη συζήτηση αναφέρθηκε ε, η πράσινη διαμόρφωση του συστήματος μεταφορών από την, την πρώτη ομιλήτρια. Νομίζω ότι αυτό είναι σωστό. Θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι επιλέγεται ο πιο φτηνός ε, τρόπος, τελικά θα προτιμηθεί η οδική μεταφορά, αλλά νομίζω ότι εμείς θα πρέπει να επιλέξουμε τις σιδηροδρομικές ε, μεταφορές και αυτές να προωθήσουμε. Θα πρέπει να είμαστε αποδοτικοί. Νομίζω ότι μπορούμε να ενταχθούμε από τη συζήτηση που διεξήχθη πριν από 8 χρόνια στην Ολλανδία. Είχε, είχε ανακηρυχθεί μία, ένα σύστημα επιβολής ε, τελών. Η συζήτηση αυτή δεν συνεχίστηκε. Δεν θα πρέπει να επιλέγουμε δηλαδή τον πιο φτηνό τρόπο μεταφορών στην Ευρώπη. Θα πρέπει να επιλέγουμε τον πιο φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο και επίσης για να αποτρέπεται η μεταφορά, να μην υπάρχουν μεταφορές όπου δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν. Έγινε μία συζήτηση για το κατά πόσο θα πρέπει να γίνει σύνδεση μεταξύ της επιβάρυνσης των φορτηγών και της επιβάρυνσης των δυτικών όχημάτων. Από τεχνικής άποψης είναι ενδιαφέρον το θέμα αυτό αλλά πρόκειται για ένα θέμα που συζητιέται και εθνικά στα κράτη-μέλη. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ρυθμιστεί αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γίνονται διάφορε συζητήσει για ευρωπαϊκά σήματα τελών κυκλοφορία, ηλεκτρονικά διόδια κτλ. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να προσθέσουμε κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα αν είναι τόσο δύσκολε οι συζητήσει σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε, να προσπαθήσουμε να συντονίσουμε και να συνδυάσουμε την τεχνολογία μας για να μπορούμε να πληρώνουμε και σε άλλη χώρα τα συστήματα, τα συστήματα τα ίδια. Αυτό μας απασχολεί εδώ και χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τέλος. για την προσέγγιση του εισηγητή. Νομίζω ότι μας δίνει μια ευρία προσέγγιση ο κύριος Ελκαντράου και πολλές λύσεις. Αλλά ελπίζω αν τελικά επιτευχθούν ε, συμβιβασμοί να μην απομακρυνθούμε υπερβολικά πολύ από την στοχοθέτηση και να μην παραμείνει το, το πρόβλημα χωρίς λύσεις είπε ο εισηγητής, ε, χρησιμοποίησε τη λέξη προσέγγιση. Ελπίζω να παραμείνουμε στο δυνατό πιο κοντά ένα στον άλλο. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχουμε 7 συναδέλφους που έχουν το λόγο. Σίγουρα πρέπει να ακούσουμε και την Επιτροπή και πρέπει να δώσουμε στον κύριο Αλκαντράδη το χρόνο για να απαντήσει και μετά θα συζητήσουμε την έκθεση για Ζεμπόφσκι. Άρα τι να, τι να κάνουμε. Τι να πω. Βεβαίως δεν μπορώ να στερήσω το λόγο από τους συναδέλφους. Σας παρακαλώ όμως, όμως επιλέξτε ένα σημείο στο οποίο θέλετε να αναφερθείτε και πολύ γρήγορα ε, τονίστε αυτό το σημείο. Δύο λεπτά. Κύριε Ράκ, πρώτα απ' όλα έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι καλό το γεγονός ότι ο εισηγητής μας προσπάθησε να λάβει στα σοβαρά τις ε, γραμμές που είχαμε δώσει από το Κοινοβούλιο. Προσπαθεί να συγκεντρώσει μεγάλη πλειοψηφία για τις θέσεις του για να καταλήξει σε ένα συνεκτικό κείμενο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις μετέπειτα συζητήσεις με το Συμβούλιο. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα, το ανέφερα άλλωστε και σήμερα, για τις ε, ορεινές περιοχές που δεν αναφέρονται γιατί δεν έχει νόημα να υπολογίζεται ένα κόστος το οποίο εκ των υστέρων θα επιστραφεί. Ελπίζω λοιπόν να διατηρηθεί η τροπολογία υπαριθμών 20. Για τη συμφόρηση μια λέξη να πω δύο λόγια. Αν ληφθούν ε, μέτρα για τη συμφόρηση θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποτραπούν, να αποτραπεί η φορολογία της συμφόρησης. Σκοπός μας να μην είναι να τιμωρήσουμε, να εισπράξουμε, αλλά σκοπός του μέτρου θα πρέπει να είναι να βρεθούν σωστές λύσεις. Λάκτφριντ. για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι και εγώ πολύ σύντομος. Θα ήθελα να πω εξ αρχής, να πω ποιο είναι το θέμα. Η όλη οικονομία των μεταφορών κάθε χρόνο προκαλεί κόστος 150 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά 150 δισεκατομμύρια ευρώ πληρώνει μόνο 50 δισεκατομμύρια ευρώ φορολογίες και επιβαρύνσεις. Από τα 50 δισεκατομμύρια αυτά τα 16 μόνο μένουν. Αν το σύστημα όπως το προτείνει ο εισηγητής εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη-μέλη τα διόδια αυτά, τα τελευταία 16 δισεκατομμύρια θα τετραπλασιαστούν, θα πενταπλασιαστούν επειδή είμαι νομικός. Δεν θέλω να σας πω πόσο είναι το τετραπλάσιο του 16, αλλά σε σύγκριση με τα 150 δισεκατομμύρια δεν είναι πάρα πολλά. Αυτό μόνο ήθελα να αναφέρω το κόστος αυτό δεν πρέπει πάντα να προδιαγράφεται. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να αποτρέπει τη δημιουργία του κόστους αυτού. Αυτός είναι ο στόχος. Τουλάχιστον ε, αν βελτιώνονται πάντα οι μεταφορές των ε, φορτηγών. Άλλωστε να μην ξεχνάμε ότι μόνο κατά 45% είναι γεμάτα τα φορτηγά, άρα μάλλον είναι υπερβολικά φτηνά και αν το διοργανώσουμε καλύτερα το σύστημα, θα βοηθήσουμε την οικονομία, τα φορτηγά, την ατμόσφαιρα και να κλείσω λέγοντας ότι συμφωνώ εν μέρη με αυτά που ακούσαμε. Θα ήθελα όμως να πω, η συνάδελφος Βόρτμαν Κόλ ανέφερε τον μεγάλο αριθμό των τροπολογιών που έχουν υποβληθεί και θεωρεί ότι αυτό αποτελεί κριτική στο έργο του εισηγητή. Και εγώ υπέβαλα δύο-τρεις ε, τροπολογίες για την οδηγία αυτή. Και αυτός ο τεράστιος ε, αριθμός ε, τροπολογιών δεν προέρχεται από μία και μόνο κατεύθυνση. Προέρχεται από αυτούς που θεωρούν, για παράδειγμα, ότι είναι ευρύ το πεδίο, ότι δεν είναι ευρύ το πεδίο, αλλά νομίζω ότι καταδεικνύουν τελικά ότι ο εισηγητής κινήθηκε προς τη σωστή κατεύθυνση και έκανε σωστό έργο. Ελπίζω να συμφωνήσουν μαζί μου οι συνάδελφοι. Και νομίζω ότι θα καταφέρουμε πάρα πολλά στον τομέα των μεταφορών αν τελικά περάσουν οι συμβιβαστικές τροπολογίες. <coughs> Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ονέχταν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με όλο το σεβασμό, βεβαίω και θα κρατήσω τα δύο λεπτά. Α, γιατί εγώ μια πτυχή θέλω να τονίσω αυτή τη πρόταση. Η πρόθεση είναι καλή, αλλά η εκτέλεση θα μπορούσε να είναι φρικτή. Αυτό με φοβίζει πρέπει να συνδεθεί με μία σειρά από παράγοντες. Διότι δυστυχώς, παρόλο που προσπαθούμε να το πράξουμε ε, και να το πετύχουμε, η Ευρώπη δεν είναι η, δεν βρίσκεται, στην Ευρώπη δεν βρίσκονται όλοι στην διαμήρα. Εγώ έρχομαι από την Ιρλανδία και πιστεύω ότι αυτή η πρόταση θα ε, ε, ε, είναι εις βάρος μας. Εμείς είμαστε μια μικρή εξαγωγική χώρα. Τι θα κάνουμε, πώς θα φτάσουμε στην αγορά της Ευρώπης. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό, να είστε ε, δίκαιοι και να κρατήσετε τις αναλογίες. Βεβαίως, κρατήστε τις προθέσεις, αλλά εκτελέστε τις προθέσεις σας με ισότιμο και δίκαιο τρόπο. Διαφορετικά, μην τις εκτελέσετε καθόλου. Κύριος Κράμερ, ένα λεπτό μόνο, γιατί κύριος Λίχτεμπεργκερ μας πήρε πολλή ώρα. Sorry, sorry, you're right. She used, she used a lot of time. <laughs> she used a lot of time. She used. <laughs> okay. Ο κύριος Λάιχτφριντ ανέφερε τα αριθμητικά στοιχεία. Γιατί μιλάμε. Μιλάμε για τη μείωση για των φορολογικών προνομίων. Να τα ακούσει και ο Γιατζεμπόφσκι. Ακόμα και αν έχετε αντίρρηση, είναι τεκμηριωμένα τα γεγονότα αυτά. Για τα τρένα, για κάθε ατμομηχανή, έχουμε συμφωνήσει να υπάρχουν διόδια για το συντηροδρόμο. Παντού στην Ευρώπη και στις οδούς δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς μπορούμε να δεχόμαστε αυτή την αδικία. Αυτά τα προνόμια θα πρέπει να καταργηθούν. Είσαστε δεκάδες χιλιόμετρα πίσω. Αν δεν, καταλάβουμε, να, αν καταφέρουμε να πετύχουμε αυτά τα μικρά βήματα, αυτούς τους μικρούς συμβιβασμού, γιατί οι οδικές κυκλοφορίες, οι οδικές μεταφορές οφείλονται για το 30% των εκπομπών αερίων δεν θα μπορέσουμε να σώσουμε το κλίμα και τις επερχόμενες γενιές. Δεν θα πρέπει να τα αποδυναμώνουμε όλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, ε, δεν θέλω να επικρίνω καθόλου ε, τον κύριο Κατράου σε προσωπικό επίπεδο. Ε, ε, η εργασία του είναι πάρα πολύ καλή, αλλά η πρόταση πιστεύω ότι είναι α, δεν είναι σκόπιμη. Ε, οι 530 τροπολογίες ακριβώς δείχνουν ε, το, που, το πώς ε, αισθάνονται και, αισθάνονται και τα μέλη της Επιτροπής αλλά και οι εμπλεκόμενοι εταίροι. Υπάρχει λοιπόν ε, δυσαρέσκεια ανεξάρτητα με την κατεύθυνση στην οποία ε, ε κινούνται οι τροπολογίες. Κοιτάξτε, πρότεινα ένα νέο, εκτιμώντας μια νέα αιτιολογική σκέψη που αναφέρεται στο εξή. Λαμβάνοντα υπόψη την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη, λαμβάνοντα υπόψη συγκεκριμένα την οικονομική κατάσταση του κλάδου των μεταφορών, θα πρέπει να ε, σκεφτούμε ε, την πρόταση αυτή ε, και να, με, μια σοβαρότητα επί της ουσίας και να παρατείνουμε τις, τις προθεσμίες. κοιτάξτε, εγώ υπέβαλα περίπου 30 τροπολογίες, όχι μόνο, μου, αλλά και με άλλους συναδέλφους που έχουν παρόμοιες ανησυχίες. Μα σε δύο λεπτά δεν μπορούμε τώρα να κάνουμε μια ανάλυση των τροπολογιών. Λυπάμαι που δεν έχουμε το χρόνο. Θα έπρεπε το θέμα αυτό να έχουμε περισσότερο χρόνο. Το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, λοιπόν, εντάξει, τηλεγραφικά θα μιλήσω, Πρόεδρε. Πρώτον, ε, όσον αφορά το τέλος για τη συμφόρηση, διαφωνούμε, σαφώ, σαφώς γιατί τα φορτηγά δεν είναι τα μόνα που ε, προκαλούν συμφόρηση. Πεδίο εφαρμογή. Η θέση μα όσον αφορά το σημείο αυτό ε, επικεντρώνεται στο ότι ε, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τελών Κυκλοφορία θα πρέπει να επιβάλλεται μόνο στου δρόμου που εντάσσονται στο ευρωπαϊκό, στα ευρωπαϊκά δίκτυα. Όσον αφορά το σημείο 2, έχουμε υποβάλει μια σειρά από έτσι ώστε να γίνει πιο συγκεκριμένο. Τα έσοδα. Στόχο πρέπει να είναι όλα τα έσοδα που προέρχονται από, αυτούς, από αυτά τα τέλη να ε, αφορούν, να, να, χρησιμοποιηθούν στις μεταφορές με ιδιαίτερη ε, προσοχή ε, στις οδούς. Όσον αφορά την 31η Δεκάτου 2013, για να υποβάλει πρόταση η Επιτροπή για το εξωτερικό κόστος, να, δεν θέλουμε να συμπεριληφθεί αυτό και η πρόταση συμπεριλάβει και άλλες κατηγορίες οχημάτων. Όσον αφορά τα μέγιστα όρια, προτείνει ο εισηγητής σε μια συμβαστική πρόταση ε, πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, λέει ο πρόεδρο. Ένα δευτερόλεπτο, πρόεδρε, ένα δευτερόλεπτο. Μα δεν έχει νόημα, λέει ο πρόεδρο. Κύριε πρόεδρε, κοιτάξτε. Με όλο το σεβασμό. Δεν είναι τρόπο αυτό ε, ε αντιμετώπιση. Ε, αυτά ήθελα να πω, πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι. Λέει Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά επιτρέψτε μου. Κοιτάξτε, πολλά από αυτά τα οποία είπατε τα, τα ανέφερε και ο εκπρόσωπος της ομάδας σας. Κοιτάξτε, έχουμε ξεπεράσει το, ε, τα χρονικά όρια ε, κατά ένα τέταρτο. Δεν φταίνε οι τελευταίοι συνάδελφοι που πήραν το λόγο, αλλά τι να σας πω. Ε, Κοιτάξτε, ε, ο, ο εκπρόσωπο τη ομάδα ε, αναφέρεται γενικά στο θέμα, συνοψίζει και εσείς αναφέρετε ένα συγκεκριμένο θέμα. Σας ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να δώσω να, να κάνω διακριτική μεταχείριση. Διαφορετικά, τι να σα πω. Μα κοιτάξτε, Διαφορετικά κανείς δεν θα καταλάβει ε, γιατί υποβάλλουμε τις τροπολογίες. Ωραία, ωραία, λέει ο πρόεδρος. Τότε πιστεύετε ότι οι εκπρόσωποι ε, τη ομάδα δεν αναφέρονται καθόλου στις τροπολογίε. Ή πείτε το εσείς, ή α το είναι οι εκπρόσωποι των ομάδων. Μα λέτε ίδια και τα ίδια συνέχεια. Δεν έχουμε χρόνο. Σίμψον. Θα είμαι σύντομο. Ουσιαστικά, βλέποντας ε, την έκθεση, ο εισηγητής δούλεψε πολύ και προσπάθησε να συμμετέχουν όλοι. Δεν μπορούμε όμως να είμαστε υπέρ των πράσινων μεταφορών και από την άλλη πλευρά να θέλουμε να παραμείνει το status quo. Από τη μία πλευρά να λέμε ότι ο εισηγητής έκανε καλή δουλειά και από την άλλη να λέμε ότι δεν θα συμφωνήσουμε με τους συμβιβασμούς. Και δεν μπορούμε να λέμε για ένα σωρό πράγματα ας το ξεχάσουμε, γιατί τότε δεν θα καταλήξουμε ποτέ σε κάποια πρόοδο. Πώς νομίζετε ότι είχαμε και στη συμφωνία στην ασφάλεια των ε, θαλάσσιων μεταφορών. Βεβαίως ε, μπορούμε να έχουμε διαφωνίες με τον εισηγητή. Το είχαμε δει και με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και με τις λιμενικές υπηρεσίες και εκεί είχαμε τον συντονιστή σας ως συζητητή και διαφωνούσαμε, αλλά αυτό δεν σήμαινε ότι επικρίναμε το έργο του, απλά σήμαινε ότι ενδιαφέρονταν οι ευρωβουλευτές για το θέμα ιδιαίτερα. Εγώ νομίζω ότι ο εισηγητής βρίσκει ένα συμβιβασμό μεταξύ αυτών που δεν θέλουν να γίνει τίποτα και αυτών που θέλουν να γίνουν όσο το δυνατόν περισσότερα. Και είναι αλήθεια ότι θα χρειαστεί τη σοφία του Σολομώντα και τη διπλωματική δυνότητα των Ηνωμένων Εθνών. Καλή τύχη λοιπόν στον εισηγητή. Κοιτάξτε, πρέπει να αποφασίσουμε κατά πόσον θα βρούμε κάποιο συμβασμό ή όχι. Ε, Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το σημείο από το οποίο ξεκινάμε. Δεν είμαστε ακόμα εκεί πάντω. Τελευταία παρέμβαση ο κύριο Φερνάντε. Eh, ε, πρόεδρε, παρακολούθησα πολύ ε, προσεκτικά την όλη διαδικασία και νομίζω ότι και ο εισηγητής άκουσε όλους αυτούς που πρότειναν τροπολογία. Αλλά είναι αλήθεια ότι στους συμβασμούς καταλήγουμε στο τέλος της διαδικασίας. Και Γι' αυτό ε, παίρνω και εγώ το λόγο, γιατί αναφέρθηκαν διάφορε στοιχείες που δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Γι' αυτό και τα θέματα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. για να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό με έναν τρόπο που, που να είναι και κατανοητός ε, από τους Ευρωπαίους πολίτες. Τηλεγραφικά, όσον αφορά τα δίκτυα. Εγώ υποστηρίζω τα δίκτυα και πιστεύω ότι θα πρέπει ε, να ε, επεκταθούμε και σε άλλα δίκτυα. Αλλά ας περιμένουμε τώρα να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα της εφαρμογής. Στη συνέχεια πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε απαντήσεις συγκεκριμένες και να λάβουμε υπόψη τους διάφορους τρόπους μεταφοράς. Δεν μπορούμε δεν μπορούμε να ε, προβαίνουμε στη διακριτική μεταχείριση. Τώρα, ε, όσον αφορά το earmarking, να, να το περιορίσουμε στις οδικές μεταφορές. Και κοιτάξτε, όσον αφορά την αξιολόγηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Όχι μόνο για να δούμε σε τι αποτελέσματα καταλήξαμε, και κατά πόσο πετύχαμε τους στόχους, πράγμα το οποίο είναι απόλυτα σεβαστό, αλλά ταυτόχρονα πιστεύω ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα αξιολόγησης για να ανοίξουμε και άλλες πόρτες, για να ανοίξουμε και άλλες οδούς. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να φερθούμε σε αυτό το είδος της αξιολόγησης. Ε, αυτό ήθελα να πω πρόεδρε σε αυτό το στάδιο. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ε, λοιπόν, ε, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Γιατζερμπόφσκι. Πρόεδρε, ο κύριο Σίμψο είναι μάστρος στο θέατρο. Αλλά μα λέει ανοησίε. Η αντίθεση ότι μια ομάδα δεν θέλει να κάνει τίποτα και όλες οι υπόλοιπες θέλουν να δράσουν είναι εσφαλμένη. Να σας πω λοιπόν ότι υπάρχει και μία αντικειμενική απόφαση. Για παράδειγμα για το κόστος της συμφόρησης. Η συμφόρηση προκαλείται από κράτη-μέλη που δεν αναπτύσσουν αντικειμενικές υποδομές. Δηλαδή το κράτος μέλος προ, προκαλεί τη συμφόρηση και ζητά δηλαδή χρήματα τελικά μόνο από τα φορτηγά και όχι από τα ιδιωτικά οχήματα που προκαλούν το 80% της συμφόρησης. Υπάρχει και η δικημενική πλευρά. Κοιτάξτε, ε, είναι ξεκάθαρο το θέμα, αλλά νομίζω, ότι το κλίμα είναι καλό έτσι, μην το ξεχνάμε. Ε, θα, θα καταφέρουμε να έχουμε συμβασμούς, μην ανησυχείτε. Κοιτάξτε, ε, εντάξει, τα γνωρίζουμε όλα αυτή τη στιγμή στι διαπραγματεύσει ε, ο καθένα προσπαθεί να πετύχει όσο το περισσότερα. Αλλά θα υπάρξουν συμβασμοί, μην ανησυχείτε. Το πρόβλημα να δούμε τι θα γίνει και με την άλλη επιτροπή. Θα μα βοηθήσει. Euh, euh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αισθάνομαι λίγο θύμα της ε, πολύπλοκης αυτής συζήτησης γιατί θα μιλήσω στο τέλος αλλά θα προσπαθήσω και εγώ να επικεντρωθώ στα βασικά. Καταρχάς να πω ότι η πρόταση είναι κομμάτι μιας συνολικής στρατηγικής αποτελεί απάντηση σε ένα έτοιμο του Κοινοβουλίου γιατί θυμάστε την ε, συμβιβαστική πρόταση που είχε γίνει τέλη 2005-2006 και η πρόταση δεν είναι φόρος απλά αλλά είναι μέτρο της ε, πολιτικής μεταφορών. Επειδή είναι τόσο σημαντικές οι οδικές μεταφορές, πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο και στην πολιτική που ασχολείται με τη βιωσιμότητα των μεταφορών. Και για όσους αντιτίθενται θα ήθελα να μιλήσω και για το εξής παράδοξο. Είτε οι αντίθετοι είναι, προέρχονται από περιφερειακές χώρες είτε άλλοι ευρωβουλευτές. Αρκετά κράτη-μέλη ήδη σκέφτονται ή εφαρμόζουν τρόπους κοστολόγησης των υποδομών πέρα από αυτά που προβλέπει η υπάρχουσα οδηγία. Οπότε είναι προς το συμφέρον το δικό μας αλλά και του επαγγέλματος να υπάρξει ένα κοινοτικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει την ίση μεταχείριση, τη διαφάνεια και την ύπαρξη βιώσιμης ε, και ισότιμου ανταγωνισμού. Και εδώ να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για το τεράστιο έργο του, αλλά και όλους τους σκιώδεις εισηγητές που συνεργάστηκαν ο καθένας με τις ιδέες του και τις ευαισθησίες του, αλλά όλοι συνεισέφεραν στο συλλογικό έργο δύο θέματα, συμφόρηση και earmarking. Όσον αφορά τη συμφόρηση, κατανοούμε το πρόβλημα που προκύπτει αν πούμε ότι η πρόταση χτυπάει ορισμένα μόνο από τα αυτοκίνητα που συνεισφέρουν στην κυκλοφοριακή συμφόρηση. Υπάρχουν όμως λόγοι πίσω από αυτό. πρέπει να μην ξεχνάμε ορισμένες ουσιαστικές συνιστώσεις. Και πρέπει να θυμόμαστε ότι η αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης σημαίνει και μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα χωρίς να προσθέσουμε επιπλέον φορολογία για το διοξίδιο του άνθρακα στην Ευρωβινιέτα. θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε εξοικονόμηση καυσίμων και γενικά σε διάφορες ε, οικονομίες ε, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν επιπλέον όπως είπα και στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Βεβαίως έχουμε και την άλλη συνιστόσα της κυκλοφοριακής ε, συμφόρησης, τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης. Εδώ έχουμε ένα παράδοξο μπροστά μας. Τα κράτη-μέλη είναι απολύτως ελεύθερα να χρεώσουν τα γιοταχή στη χώρα τους για αυτό, αλλά δεν μπορούν να το κάνουν στην περίπτωση των βαρέων οχημάτων γιατί ισχύει η οδηγία για την Ευρωβινιέτα. Έχουμε λοιπόν μία άνηση μεταχείριση εδώ. και ένα σχέδιο δράσης βεβαίως δεν θα μπορούσε να επιλύσει το πρόβλημα της κυκλοφοριακής ε, συμφόρησης, ε, περισσότερη γραφειοκρατία θα σήμαινε μάλλον. Θα μπορούσαμε όμως να έχουμε ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα συνέδεε το θέμα με τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης. Και περνάω τώρα στο θέμα του earmarking. Όλοι μιλάνε γι' αυτό και είναι και η δική μας προσέγγιση. Όντως έχουμε πει ότι η Ευρωβινιέτα δεν είναι απλά φορολογία, είναι μέτρο της πολιτικής μεταφορών και ως τέτοιο πρέπει να το δούμε και τώρα. Βρισκόμενοι αυτή την περίοδο σε οικονομική κρίση, θεωρούμε ότι ο τρόπος να την αποφύγουμε είναι μέσω και των επενδύσεων στις υποδομές. Και για να γίνει αυτό χρειάζονται πόροι. Γιατί αν δεν υπάρχουν χρήματα, δεν λαμβάνει χρήματα από τους φορολογούμενους το κράτος δεν θα μπορέσει να δημιουργήσει νέες υποδομές με κάλυψη και του εσωτερικού και του εξωτερικού κόστους. Επειδή βλέπω ότι όλοι σας είστε υπέρ του earmarking, θεωρώ ότι είναι αντιφατικό. Από τη μία πλευρά <laughs> να ζητάμε earmarking, από την άλλη πλευρά όμως να προσπαθούμε να αδειάσουμε την οδηγία από ορισμένε βασικές συνιστώσεις της, όπως αυτή που αφορά την συμφόρηση, γιατί μόνο μέσα από τέτοιους σημαντικούς πόρους θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο για να επιτύχουμε μια βιώσιμη πολιτική μεταφορών και μια αύξηση των επενδύσεων στις μεταφορές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος θα είμαι σύντομος, Πρόεδρε. Έχετε το δικαίωμα να πείτε ότι θα το σκεφτείτε. Ναι, φυσικά και θα το σκεφτώ, αλλά θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι θεωρώ ότι στο Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να διαμορφώσουμε μια πολύ σαφή θέση. Δεν θα πρέπει να κάτσουμε να ανησυχούμε τι θα δεχτεί το Συμβούλιο και τι όχι. Πρόκειται δικά μας θέματα θα καταρτήσουμε νομοθεσία για ένα κλάδο στον οποίο υστερούμε για το μέλλον. Σας εγγυώμαι ότι και εγώ προσωπικά θα επενδύσω πολλά, αλλά θεωρώ ότι η υποστήριξη την οποία θα μπορούσαν να λάβουν οι συμβιβαστικέ προτάσεις δεν θα προκύψει σε περίπτωση που δεν θα προκύψει συμφωνία με το Συμβούλιο. Υπάρχει λοιπόν έντονη πίεση για να μην υποχωρήσουμε σε κάποια θέματα. Σε αυτά θα περιοριστώ συνάδελφοι. Τις επόμενες εβδομάδες ε, θα ξαναχτενίσουμε κάποιες ε, προτάσεις μου. Καταλαβαίνετε δεν θα καταφέρουμε να ικανοποιήσουμε τους πάντες 100% και να τους κάνουμε να υποστηρίξουν την ε, πρόταση αυτή γιατί υπάρχει υπερβολική διάσταση απόψεων αλλά νομίζω ότι με καλή θέληση από όλου, με αρκετή ευελιξία θα καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε αρκετή πλειοψηφία για να υποστηρίξει κάποιες βασικές ιδέες. Ευχαριστώ. Bene. Πολύ ωραία. Με μισή ώρα καθυστέρηση περνάμε σε ένα θέμα όχι πολύ διαφορετικό, που έχει να κάνει με το θέμα του κυρίου Γιαζερβόφσκι. Αγαπητοί φίλοι, ήθελα να ήμουν στο γραφείο μου να ακούω και τι λέει ο Ομπάμα στην ορκομοσία του. Γι' αυτό θα είμαι σύντομος για να προλάβω τουλάχιστον το δεύτερο μέρος. Και νομίζω ότι η στοχοθέτησή μου είναι η ίδια με αυτή του Ελκαντράουι. Θα προσπαθήσω για την ε, έκθεσή μου να συγκεντρώσω μια αρκετή πλειοψηφία, αν θέλετε, πίσω από κάποιες αρχές. Η αρχική μου έκθεση ήταν αρκετά προκλητική ίσως για κάποιους, αλλά είμαι και εγώ παλαιός νομικός, βλέπετε. Υπάρχει διαφορά μεταξύ ε, του προκλητικού και του θεατρικού. Αλλά ας αφήσουμε κατά μέρος τις γλωσσικές αυτές ε, λεπτομέρειες. Διατύπωσα 12 τροπολογίες για να δούμε, για να δημορφωθεί πλειοψηφία. Συμπεριέλαβα στις συμβαστικές τροπολογίες σειρά σχολείων των συναδέλφων. Συμπεριέλαβα και τις προτάσεις του Ελκαντράου για το Ευρωπαϊκό Σήμα Τελειών Μεταφοράς Κυκλοφορίας στην παράγραφο 7, 9, 11. Τροποποίησα σαφώς τη διατύπωση. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε πλειοψηφία υπέρ των προτάσεων αυτών εδώ στην Επιτροπή Μεταφορών. Είναι σημαντικό πιστεύω επί της αρχής για ένα γενικό σύστημα να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε ένα δίκαιο σύστημα. Αυτό νομίζω μας βρίσκει σύμφωνους. Ε, συμφωνήσαμε άλλωστε ότι δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό το Ευρωπαϊκό Σήμα Τελών Κυκλοφορίας για όλες τις ε, χώρες. Αλλά σε ό,τι αφορά θέματα αρχής στην έκθεσή μου θα πρέπει να τονίσουμε ότι αν θέλουμε να διαμορφώσουμε τις μεταφορές με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ίδιες αρχές σε όλα τα κράτη-μέλη. Δεν μπορεί να έρχεται και να μας λέει η Μάλτα ότι «Α, εμένα δεν με νοιάζουν οι διατάξεις σας γιατί είμαι νησί». Γι' αυτό λοιπόν ε, και συμπεριέλαβα τις αλλαγές που συμπεριέλαβα. Προτείνω να μην υπερψηφιστούν κάποιες τροπολογίες στον κατάλογο ψηφοφοριών. Ψηφο... που αναφέρονται σε θέματα κλίματος, γιατί αυτά συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο του κλίματος που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο. Για παράδειγμα το 20% μέχρι το 2020 και όλα αυτά. Όλα αυτά έμα ε, τα συζητήσαμε και τα αποφασίσαμε ήδη. 17 Δεκεμβρίου νομίζω ήταν στο πακέτο για το περιβάλλον. Δεν έχει νόημα θεωρώ να τα επαναλαμβάνω στην έκθεσή μου. Γι' αυτό να ζητήσω την κατανόηση των συναδέλφων και να με συγχωρέσουν που δεν μπορώ να συμφωνήσω με τις τροπολογίες αυτές. Γιατί αν το Κοινοβούλιο έχει πει κάτι και έχουμε πει πολύ σημαντικά πράγματα το Κοινοβούλιο στο πακέτο για το κλίμα με συντριπτική πλειοψηφία, ε, δεν χρειάζεται να τα ε, επαναλαμβάνουμε κάθε φορά σε κάθε διαδικασία. Γι' αυτό ελπίζω οι συνάδελφοι να μπορέσουν ε, να αποτεχτούν τι συμβιβαστικέ προτάσει. Ε, κάποιοι από την ομάδα μου μου λένε πώ μπορεί να φτάνει μέχρι το σημείο αυτό. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει η αρχή που διέπει την έκθεση να είναι η διαμόρφωση των μεταφορών με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Και ελπίζω, σε αυτό το πνεύμα επιβάλλα και τις τροπολογίε μου, ελπίζω να σας βρουν σύμφωνος. Ο ε, κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι και εγώ σύντομος, γιατί και εγώ θέλω να ακούσω το δεύτερο ήμιση της ομιλίας του Ομπάμα. Λέει ο γιατί ότι ήταν πολύ προκλητική του πρώτη σου. Και εγώ να σας πω ότι και εγώ και η ομάδα μου εκτιμούμε τις προσπάθειες που έγιναν για να μας προσεγγίσετε και για να καταλήξουμε σε κάποιες συμβαστικές προτάσεις. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για το έργο σας αυτό φυσικά παραμένετε εξαιρετικά κριτικός, επικριτικός και νομίζω ότι αυτό είναι λογικό. για να καταλήξουμε εκεί που θέλουμε σε ένα βιώσιμο σύστημα για όλα τα είδη μεταφορών. Άρα, λάβαμε γνώση των συμβαστικών προτάσεών σας και σε μεγάλο βαθμό μπορούμε να τις υποστηρίξουμε δεν προβλέπω δηλαδή να υπάρχουν ε, σωματικά προβλήματα. Φυσικά έχουμε και άλλες ε, και έχουμε και κάποιες τροπολογίες που θα θέλαμε να τύχουν υποστηρίξεις, αλλά αυτό θα αποδειχτεί στην ψηφοφορία αν θα υπερψηφιστούν ή όχι. Πάντως, συνάδελφε, για Ζεμπόφσκι είναι, σημαντικό, είναι πραγματικά εκπληκτικό το πόσο, πόση απόσταση καλύψατε. Κύριε Στέρξ, ε, ευχαριστώ. Δεν ε, υπέβαλα τροπολογίε, οπότε ε, δεν με αφορούν άμεσα οι συμβιβαστικέ προτάσει του κύριου Ζεμπόφσκι. Θα ήθελα να ρωτήσω και του δύο συναδέλφου να του πω ότι οι δύο εισηγήσει, οι δύο εκθέσει δεν μπορούν να είναι αντιφατικέ. Θα πρέπει να υπάρχει ένα συντονισμό. για να είναι σαφές το τι επιθυμεί και η Επιτροπή Μεταφορών. Και σε ό,τι αφορά τις συμβαστικέ προτάσεις για τη δική σας έκθεση, ίσως θα πρέπει να τροποποιηθούν, θα πρέπει να προσαρμοστούν οι μεν στις δε. Κυρία Λίχτενμπέργκερ, σας ευχαριστώ. Και έχετε δίκιο κύριε συνάδελφε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία του Ομπάμα. Και σε αντίθεση με αυτά που μας είπατε εσείς, δίνουν και ελπίδα για το μέλλον. Τώρα το κατά πόσο θα μπορέσει ο Πρόεδρος να πραγματοποιήσει την ελπίδα αυτή, ε, αυτό θα το αποδείξει το μέλλον σαφέστατα. Αυτό που βλέπω εδώ, πάντως μπροστά μου, δεν μου δίνει καμία μεγάλη ελπίδα, επειδή σε πρώτη γραμμή ουσιαστικά ε, επικρίνεται το οτιδήποτε θα μπορούσε να προσωμιάσει συγκεκριμένο μέτρο. Στην πραγματικότητα θέλετε να περιμένουμε λίγο ακόμα, να περιοριστούμε στην αναμονή αυτή, να θέσουμε το στόχο, να το κοιτάξουμε κάποια χρόνια το στόχο αυτό, να σκεφτούμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Αυτά δεν μου αρκούν, γιατί η κατάσταση είναι δραματική και δεν επιτρέπει τέτοια χρονοτριβή. Θα ήθελα λοιπόν πιο συγκεκριμένα στοιχεία να συμπεριληφθούν. Πέρα από την κριτική που περιλαμβάνεται στην έκθεσή σας. Εγώ δεν είμαι ικανοποιημένη. Δεν με ικανοποιούν αυτά που μας ε, προτείνετε, αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα περιμένετε και τίποτα διαφορετικό από εμένα. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, δίστανται οι απόψεις για το τι είναι σημαντικό για την ευρωπαϊκή πολιτική. Το όφελος για το ευρύ ή για συγκεκριμένους κλάδους. Έτσι έχει ζωή, τι να κάνουμε, λαμβάνω γνώση της κατάστασης, ε, υπάρχει διάσταση απόψεων, αλλά μακάρι να κάνετε και κάποια στιγμή ένα βήμα προς τα εμάς. Λοιπόν, δεν βλέπω κανείς άλλο θέλει το λόγο να ζητήσω από την Επιτροπή να σχολιάσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από πλευράς Επιτροπής εκτιμούμε ιδιαίτερα τις τροπολογίες και τους συμβιβασμούς που αναγνωρίζουν ότι απάντησε η Κομισιόν ακριβώς σε αυτά που ζήτησε το Κοινοβούλιο και μάλιστα έκανε ακόμη και παραπέρα γιατί εφαρμόζει την αρχή της εσωτερήκευσης του κόστους ακόμη περισσότερα. Η Κομισιόν έκανε ανάλυση αντικτύπου, πρότεινε ένα σχέδιο το οποίο βασίζεται σε κοινέ αρχές. Όπως βλέπετε στο κεφάλαιο 3 μιλάμε για το... Όχι, δεν μιλάμε για το μέσο κοινωνικό κόστος, αλλά για το εξωτερικό το marginal ε, social cost και ναι μεν ε, σε κάποια σημεία χρησιμοποίησαμε το μέσο κοινωνικό κόστος, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος χρησιμοποίησαμε το marginal cost. Και επίσης η στρατηγική αυτή αφορά όλες όλους τους τρόπους μεταφοράς, όλα τα μέσα μεταφοράς, ακριβώς όπως είχε ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην απόφαση για την Ευρωβινιέτα. Χαιρόμαστε που βλέπουμε και τροπολογίες που μας υπενθυμίζουν την ύπαρξη των τεχνικών παρατημάτων, που συνήθως τα ξεχνάμε, παρόλο που περιέχουν πολύ σημαντικά θέματα, αλλά δυστυχώς και πολύ περίπλοκα. Κρίμα που δεν μπορούμε να τα απλωστοποιήσουμε περισσότερο, αλλά είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα τα θέματα αυτά. Και θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιαζεμπόφσκι, να σκέφτεστε τον Ομπάμα. Μία μικρή παρατήρηση. Αγαπητή κυρία Λίχτενμπεργκεν, δεν είμαι ικανοποιημένο με την Κομισιόν για το 2006 και τα προηγούμενα έτη, πριν ελευθερίνει οι αποφάσει τη 2006, είχαμε ζητήσει από την Κομισιόν να μας υποβάλει σχέδια για όλους τους τρόπους μεταφορών για την εσωτερικοποίηση του εξωτερικού ε, κόστους και για πάρα πολλά δεν λάβαμε τίποτα. Μιλώντας όμως ε, για την εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους ε, ε, για όλους τους τομείς, γιατί θα έπρεπε να έχει τεράστιο έργο η Κομισιόν. Αν δεν καταφέρει λοιπόν η κομισιόν να μιλήσει για το πραγματικό κόστος και δεν το αναφέρει καν αυτό και αναφέρει ότι ναι, όλοι οι παράγοντες μεταφοράς πρέπει να καταβάλουν το πραγματικό τους κόστο και το εξωτερικό κόστος. Καταλαβαίνετε το θυμό μου, γιατί η Κομισιόν δεν έχει καταφέρει αυτό που θέλαμε από αυτήν ως τώρα και ούτε την πρόταση του Δήμα έχω δει, ούτε για την δημιουργία τις ε, πράξης του Μανχάιμ και για τις τιμές του θορύβου για τα τρένα που ενοχλούν τον πληθυσμό. Θέλουμε να κάνουμε πιο πολλά και πιο γρήγορα, αλλά όλα αυτά θα τα ψηφίσουμε στις 11 και να δούμε τι μπορούμε να προλάβουμε από τον Ομπάμα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε αύριο σε 9.